Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. E Σας καλωσορίζουμε στην ε, αίθουσα του ΕΛΚ. Σήμερα λοιπόν έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση που θα χωριστεί σε τρία τμήματα. Καταρχήν θα έχουμε την ακρόαση του Πρόεδρου της Επιτροπής, του κ. Γιούγκα, τον οποίο και καλωσορίζω θερμά. Μετά θα ακολουθήσει μια πιο σύντομη συνεδρίαση με τον Υφυπουργό Οικονομικών της ε, Πορτογαλίας και μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο της Επιτροπής για το, το, για το γεγονός ότι δέχτηκε την πρόσκληση της Επιτροπής μας χωρίς κανένα δισταγμό και ήρθε εδώ σήμερα για να του θέσει ερωτήσεις και να απαντήσει. Έχουμε ήδη συζητήσει δύο φορές με τον κύριο Μοσκοβίση και μία φορά με την κυρία Γιούροβα για την κείμενη νομολογία. Και επιπλέον η επιτροπή, η αρμόδια επιτροπή έχει μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μάλτα, στο Λουξεμβούργο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Επιπλέον ε, στην Ελβετία και στην Κύπρο και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες συνεργασίας. Οι δυνατότητες αυτές ε, δεν είναι βέβαια πάντα ικανοποιητικές και γι' αυτό κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής θα ήθελα να φέρω τρία πράγματα. Καταρχήν η πρόσβαση στα έγγραφα και εδώ διαπιστώνουμε υπάρχει μπλοκάρισμα από πλευράς ε, Κοινοβουλίου τουλάχιστον όσον αφορά Συμβουλίου, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Μπλοκάρισμα από την πλευρά του Συμβουλίου, λοιπόν, ε, γιατί αυτό δεν είναι σωστό όμως, γιατί πρόκειται για ένα διοργανικό στοιχείο. Δεύτερον, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο για την ε, συνεργασία, το πνεύμα συνεργασία που επιδεικνύει η Προεδρία τη Μάλτα. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου, υποτίθεται θα ερχόταν ε, σε εμά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει και θα δούμε πώ θα εξελιχθεί η κατάσταση. Και τρίτον, υπάρχει γενικότερα μία άρνηση διαθεσιμότητα στην Επιτροπή μα αυτό από πλευρά δικηγόρων, τραπεζιτών και γενικά πολιτικά επωνύμων. Όμω, εσεί, κύριε Γιούγκερ είστε διαφορετικό. Γι' αυτό σα ευχαριστώ και πάρα πολύ. Υπάρχουν 10 θέματα που σα έχουμε υποβάλει, που αφορούν, όπω σα είπα, στην νομοθεσία που ισχύει τώρα. Τα θέματα όμω αυτά έχουν σχέση και με προηγούμενε στρατηγικέ που ακολουθήθηκαν από πλευράς Λουξεμβούργου. Σήμερα το Λουξεμβούργο, πιστήκαμε και μόνοι μας, το Λουξεμβούργο λοιπόν είναι το δεύτερο μεγαλύτερο η μεγαλύτερη έδρα συγκέντρωση κονδυλίων στον κόσμο και είναι και η έκτη μεγαλύτερη, η έκτη χώρα όπου συγκεντρώνει τις περισσότερες τράπεζες. Ε, όταν ήσασταν αρμόδιος στο Λουξεμβούργο και εγώ τότε στη Ρινανία Παλατινάτο, πάντα πρέπει να σας πω ότι σας θαυμάζαμε και εσάς και το Λουξεμβούργο το πόσο ταχύτατα εξελίχθηκε στο να καταλάβει αυτή τη θέση που σας περιέγραψα. Σήμερα, και το λέω αυτής εξ αρχής, ε, σας το λέω γιατί σήμερα ε, θα υπάρξουν και κάποιες ε, δημοσιεύσεις από πολιτική ομάδα και υπήρξαν και κάποιες ε, φήμες που κυκλοφόρησαν. Εμείς δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Η μελέτη που έχει γίνει τουλάχιστον έτσι διάβασα στον τύπο, δεν προσφέρει κανένα καινούριο στοιχείο. Εγώ 23 χρόνια είμαι μέλος της ΕΚΟΝ και ξέρουμε ότι πέρασαν 15 χρόνια μέχρι να θεσπιστεί η οδηγία περί έδρας και δεν ήταν το Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Ολλανδία, Αυστρία, ε, τα νησιά της Μάνχης που εκπροσωπούνται από τη Μεγάλη Βρετανία και το Λουξεμβούργο. Όλοι αυτοί εμπλέκονται στην οδηγία, όχι μόνο το Λουξεμβούργο και το λέω για να δημιουργηθούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σήμερα λοιπόν δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, απλά η Επιτροπή Έρευνας θέλει να ερευνήσει τις μεθόδους, τις ε, διαπραγματεύσεις και ενδεχομένως και το ότι θα πρέπει να πράξουν κάποιες αλλαγές στην κείμενη νομοθεσία. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε προβλέψει 10 λεπτά να μιλήσετε εσείς εν είδη Και μετά ε, θα μιλήσουν και οι συγητές μας ανά πέντε λεπτά όμως θα υπάρχει δυνατότητα έρωτα απαντήσεων. Τώρα παρακαλώ οι φωτογράφοι να κάνουν ε, λίγο χώρο για να <laughs> βλέπουν οι βουλευτές τον πρόεδρο της Επιτροπής όταν θα μιλάει. Αν θέλετε λίγο στην άκρη. <coughs> Σας ευχαριστούμε λοιπόν για άλλη μια φορα Ζαν Κλοντ, έχει το λόγο. Έχει πολύ αξιότιμε πρόεδρε. Εγώ δυστυχώς ε, δεν μπορώ να μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα. Κρίμα. Γι' αυτό ε, θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του Πολτέρου για την εισαγωγή μου που δεν σημαίνει ότι δεν είμαι και προετοιμασμένος να μιλήσω αγγλικά. Κυρίε και κύριοι, βρίσκομαι εδώ μπροστά σας σήμερα διότι συμμεριζόμαστε έναν κοινό στόχο και μια κοινή βούληση για ένα διακύβημα πολύ σημαντικό που μας αφορά όλους. Η, την φορολογική δικαιοσύνη, η οποία είναι απαραίτητη ούτως ή άλλως και αυτή τη στιγμή πιο απαραίτητη από ποτέ. Αποκαλύφθηκαν οι δυσλειτουργίες καθώς και οι πρακτικές φοροαποφυγής που χρησιμοποιούν κάποιες επιχειρήσεις και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό έγινε μέσω της LuxLeaks και βεβαίως η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μα κλονίστηκε. Είναι λογικό να γανακτούν, είναι λογικό να ε, κατηγορούν αυτό το σύστημα αποφυγή τη φορολόγησης των επιχειρήσεων που παραμένει άδικο, ακατάλληλο και ε, εξαιρετικά σκοτεινό. Χρησιμοποιούν το σύστημα αυτό με πολυεθνικές επιχειρήσεις που ε, εκμεταλλεύονται τα κενά τα στο συντονισμό τις τα διαφορετικά φορολογικά καθεστώτα για να μπορέσουν να μειώσουν τη φορολόγησή του. Σύμφωνα με την εκτίμησή σα στο Κοινοβούλιο, η φορολογική απάτη αφορά 70 δισεκατομμύρια ευρώ ε, απώλεια σε φορολογικά έσοδα. Λιγότερε δηλαδή επενδύσεις, 70 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερε επενδύσεις σε κοινωνικέ υπηρεσίε Και είναι πρώτε, τα πρώτα θύματα ε, οι μικρέ επιχειρήσει. Ε, είναι 30% μεγαλύτερη φορολογική ε, το φορολογική βάση για τι μικρέ επιχειρήσει από ό,τι για τι ε, πολυεθνικέ. Είναι η κατάσταση αυτή απαράδεκτη. Διότι αυτό το σύστημα ε, πλήττει πολλού, κερδίζουν λίγοι και βεβαίω ε, πλήττεται και η αρχή τη ισοτιμίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βάλουμε τέλο λοιπόν σε αυτέ τι πρακτικέ τις αθέμητες πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πιο δίκαιοι ε, και πιο ισότιμοι. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ήδη κατά τη διάρκεια της προεκλογής εκστρατείας του 2014 στις ευρωεκλογές είχα δεσμευθεί να ακολουθήσω αυτή την οδό χωρίς κανένα δισταγμό. Είναι βούληση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου άλλωστε, την έχει εκφράσει Πολάκης και η δική μου επιτροπή από την πρώτη μέρα της εντολής της ε, είχε αναφερθεί σχετικά στις 15 Ιουλίου του 2014 ήδη είχα κάνει σχετική παρουσίαση. Όταν ήρθα στο Κοινοβούλιο στις 12 Νοεμβρίου του 2014 και όπως ε, είπα και στην Επιτροπή Ταξίου το 2015 είπαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αντιμετωπίσουμε τη φορολογική απάτη. Και σήμερα τα γεγονότα μιλάνε από μόνα τους τα αποτελέσματα. Ο Πιέρμος κοβησί, η Μάγκαριτ Βέσελ έκαναν πραγματικά πολύ καλή δουλειά. Σε δύο χρόνια εγκρίναμε φιλόδοξε μεταρρυθμίσει για να προωθήσουμε μια απλή αρχή και λογική. Πρέπει οι επιχειρήσεις να πληρώνουν τα κέρδη, τα, τους φόρους τους εκεί όπου δημιουργούν τα κέρδη τους. Ήταν μια δέσμευση της εκστρατείας μου, της προεκλογικής και θέλω να τη σεβαστώ. Κατόπιν ερευνών για τις ε, φορολογικές πρακτικές ε, ε, στην, στο Λουξεμβούργο και στις κάτω χώρες και, και άλλων πολυεθνικών στο Βέλγιο. Πήραμε και μια απόφαση κατά της Apple που θα μας οδηγήσει στο να ανακτήσουμε 13 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά κίνητρα που είχαν δοθεί. Και άλλες έρευνες είναι να εξελίξει αυτή τη στιγμή, αυτή που αφορά την Amazon ή την NGNDF e Suez, μια εταιρεία που γνωρίζουν καλά οι γαλλικές αρχές για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η αρχή θα γίνει περισσότερο σεβαστή στο μέλλον και ότι τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσουν να εγγυηθούν μια ισότιμη φορολόγηση, έχουμε θεσπίσει μια πραγματική επανάσταση. Ε, την επανάσταση της φορολογικής διαφάνειας κατά της οικονομία τη σκιάς. Προχωρούμε λοιπόν με ένταση και ταχύτητα, αλλά υπάρχουν και αντιστάσεις. Μπορέσαμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη για να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια και να δράσουμε συγκεκριμένα για να πετύχουμε τον κοινό στόχο μας μια ισότιμη φορολόγηση και αποτελεσματική. Ποιο θα μπορούσε να φανταστεί πριν από δύο χρόνια ότι μέσα σε 7 μήνες θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία για την αυτόματη αντιλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά ε, τα φορολογικά στοιχεία. Τον Ιανουάριο φέτος εγκρίθηκε αυτό, και οι πρώτες ανταλλαγές πληροφοριών θα γίνουν ήδη αυτό το καλοκαίρι. Αυτή η συμφωνία επετεύθη τον Οκτώβριο του 2015 επί Προεδρίας του Λουξεμβούργου, να το πούμε και αυτό. Πέρσι συνεχίσαμε την προσπάθεια αυτή, βάλαμε τέλος στο, στο τραπεζικό απόρριτο μια σειρά διμερείς συμφωνίες για την ε, φορολογική διαφάνεια μεταξύ των 28 κρατών μελών, το Μονακό, την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου βασιζόμαστε στο, στο BEPS, δηλαδή το πρόγραμμα του ΩΣΑ και έχουμε προτείνει μια ασπίδα κατά της φορολογικής απάτης για να αντιμετωπίσουμε τις πιο τακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις τις πιο συνηθισμένες για να αποφύγουν τους φόρους. Και πάμε παραπέρα από αυτά που προτείνει ο ΩΣΑ. Μια και οι κανόνες μας είναι δεσμευτικοί. Επίσης πήγαμε γρήγορα και πολύ μακριά σε ό,τι αφορά ε, τους κανόνες φορολόγησης ε, για τις πολυεθνικές που πρέπει να τηρούν και πρέπει να κοινοποιούν στις φορολογικές αρχές. Έχουμε επίσης προτείνει να δημοσιοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Ο κάθε πολίτης να μπορεί, δηλαδή εφόσον το επιθυμεί, να έχει πρόσβαση ε, στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων, στο ποια είναι τα κέρδη αυτά και πόσους φόρους πληρώνουν σε όλες αυτές τις χώρες. Αυτή η υποχρέωση ε, σημειώνει, αποτελεί πολύ σημαντική πρόοδο στο επίπεδο φορολογική διαφάνεια. Θέλω να πάμε ακόμα πιο μακριά. Είμαστε ακόμα στην αρχή. Η πραγματική ε, παγκόσμια σφαιρική λύση το θέμα της, για το θέμα της μεταφοράς των κερδών ε, είναι να υπάρχει μια κοινή φορολογητέα βάση για, την, για τη, φορολογία, τη φορολογία των επιχειρήσεων, για να σταματήσει να υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ εθνικών συστημάτων, σεβόμενη βέβαια το δικαίωμα της κάθε χώρας να αποφασίσει ποια θα είναι τα ποσοστά φορολόγηση των επιχειρήσεων. Γι' αυτό το λόγο, όπω και δεσμεύτηκα και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα κράτη-μέλη ε, και τι επιχειρήσει, έχουμε επαναφέρει την πρόταση του 2011 με ένα πιο απλό σύστημα και μειώνοντα το κόστο συμμόρφωσης για τι επιχειρήσει που έχουν διασνοριακέ δραστηριότητε. Αυτή η νέα εκδοχή του ειδικού φόρου κατανάλωση, του άξης μάλλον τέλο πάντων, θα εξεταστεί σε δύο στάδια. Πρώτα, η κοινή φορολογητέα βάση και όταν αυτό θα αποφασιστεί, το δεύτερο στάδιο θα έχει να κάνει με τη θέσπιση της ε, ολοκλήρωσης της ενσωμάτωσης. Αυτό θα μας επιτρέψει πολύ γρήγορα να έχουμε τα βασικά πλεονεκτήματα του άξης και για τα κρατη και για τις επιχειρήσεις πριν μπορέσουμε όλα τα πλεονεκτήματα να τα πλαισιώσουμε η άμεση απάντησή μα στο σκάνδαλο του Πάναμα, των Panama Papers είναι ότι σε λίγε εβδομάδε θα υποβάλουμε μια πρόταση για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα ε, όλους αυτούς επειδή διευκολύνουν το, τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, του διάφορου συμβούλου, συμβούλους, ε, τα διάφορα γραφεία. Επίση θα επικαιροποιήσουμε του κανόνε ΦΠΑ φέτο, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη συνοριακή απάτη που, έχουν να κάνουν, που έχει να κάνει με το ΦΠΑ επειδή πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό κατάλογο με παγκόσμιου φορολογικού παραδείσου. Θα υποβάλουμε λοιπόν ένα κοινό κατάλογο που θα μα επιτρέψει οι χώρε οι οποίε ε, δεν θέλουν να έρθουν σε διάλογο μαζί μα και δεν θέλουν να έρθουν σε συμβασμό, θα του ε, υποχρεώσουμε να ακολουθήσουν συγκεκριμένε αρχέ ορθής φορολογική διακυβέρνηση. Αυτά είναι από τα πρώτα εισαγωγικά σχόλια που ήθελα να κάνω. το Κοινοβούλιο φαντάζομαι θα υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθεια αυτή. Κάνω έκκληση προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι αλήθεια ότι τα σκάνδαλα τα οποία αποκαλύφθηκαν έχουν διευκολύνει το έργο μας, αλλά αυτή η πίεση μπορεί κάποια στιγμή να μειωθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και ε, εντατικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Ακούσαμε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, ε, τις προτάσεις της Επιτροπής και όπως είπατε και εσείς ο ίδιος, λόγω των διαφόρων σκανδάλων και των δημοσιευμάτων οι δημοσιογράφοι δημοσίευσαν αυτά τα άρθρα και με βάση τις πληροφορίες των καταγγελόντων, των whistleblowers. Θεωρούμε λοιπόν ότι η πίεση που ασκήθηκε, η πίεση αυτή ε, πραγματικά βελτίωσε την κατάσταση και επιτάχυνε τις διαδικασίες. Κατόπιν τούτου πιστεύω ότι ο στόχος μας δεν είναι τόσο τα λάθη του παρελθόντος να τα αποκαλύψουμε μετά από 20 χρόνια, αλλά να στρέψουμε το βλέμμα στο μέλλον και να μάθουμε και από εσά τι ακριβώ πρέπει να αποφύγουμε. Ε, παραδοσιακά λοιπόν έχουμε τους δύο συνεισηγητές οι οποίοι λαμβάνουν το λόγο. Ε, παρακαλώ πολύ ο πρώτος εισηγητής για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και σας χαιρετίζουμε κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Είναι μεγάλη χαρά για μας που σας έχουμε εδώ μπροστά μας στην Επιτροπή και θα ήθελα να περάσω ευθύ αμέσω στην πρώτη μου ερώτηση. Εσείς υπενηχθήκατε ότι μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες ε, των κρατών μελών είναι η μεταρρύθμιση του κώδικα διοντολογίας για, τον, για τους στην εταιρική φορολογία. Ε, εσείς επειδή ήσασταν Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου έχετε εμπειρία από πρώτο χέρι σχετικά με τον κώδικα διοντολογία. Ο στόχος της ομάδας ήταν να εντοπίσουν πολιτικές οι οποίες προκαλούν ζημιά, αλλά δυστυχώς ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Και ανταυτού προέκυψαν εμπόδια για τη διαφάνεια, για την αλλαγή και θέλουμε να γνωρίζουμε εσείς ως πρόεδρος πλέον της Επιτροπής τι θα κάνετε για να μεταρρυθμίσετε την Επιτροπή. Θα αναλάβετε την πρωτοβουλία να αξιολογήσετε τη δουλειά της τα τελευταία χρόνια γιατί αυτό μπορείτε να το κάνετε ως Επιτροπή και θα οδηγήσει αυτό σε διαφάνεια και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λύσει και το θέμα της ομοφωνίας. Ε, κατόπιν, κύριε Γιούγκερ, εσείς υπενηχθήκατε το θέμα των καταγγελόντων, τις διαρροές, όχι μόνο ε, για τα Panama Papers, αλλά και για τα Leaks και για άλλες περιπτώσεις. Η Κομισιόν λοιπόν τι προτίθεται να κάνει για να προστατεύσει καλύτερα αυτούς, αυτές τις διαρροές. Γιατί πρέπει να σας πω, είναι τραγωδία. Έχουμε τους καταγγέλλοντες οι οποίοι αποκάλυψαν τις παράνομες πράξεις της ε, λουξεμβουριανής κυβέρνησης ε, και αυτοί δικάστηκαν. Μα αυτό είναι σκάνδαλο. Θα θέλαμε λοιπόν να γνωρίζουμε κατά πόσο η Κομισιόν μπορεί να έχει ένα καλύτερο πλαίσιο για να προστατεύει δηλαδή τους ε, πληροφοριοδότες. Ε, και αυτοί ε, πρέπει να τιμώνται και όχι να τιμωρούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφε, ο πρόεδρος τώρα της Επιτροπής έχει δυνατότητα να απαντήσει για τρία λεπτά. Να πω ότι δεν έχω άμεση ε, εμπειρία για τον κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ε, δημιουργήθηκε το 1997 με δική μου πρόταση ως Πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ μαζί με μια ευρύτερη απόφαση για την οδηγία για τις καταθέσεις, τις αποταμιεύσεις μάλλον. Και φαίνεται, ε, από ό,τι είπατε, ότι δεν έχει πλήρως αποτέλεσμα. Όμως αυτό δεν είναι σωστό γιατί Έχουμε αλλάξει 421 συστήματα φορολογίας και 111 έχουν αναθεωρηθεί έτσι ώστε για να έχουμε τη σημερινή κατάσταση. Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε ε, αυτό τον κώδικα όσον αφορά στη διακυβέρνηση σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για να επιτύχουμε ακριβώς αυτό. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί ο Όμιλος και ο με τον τρόπο που ε, υπάρχει διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα τους καταγγέλλοντες, τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, νομίζω ότι η, η Κομισιόν εργάζεται επί της πρότασης πώς θα τους ε, προστατεύσουμε καλύτερα. Αυτό θα γίνει τους επόμενους ε, μήνες. Χρειάστηκα λιγότερο από τρία λεπτά. Ευχαριστώ για τα ακριβή σας ερωτήματα. Ευχαριστούμε. Είχαμε ε, προσκαλέσει τον ε, πρόεδρο της ομάδας ε, Code of Conduct. Είναι μια διακυβερνητική οργάνωση και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να κάνουμε ακρόαση από ό,τι μας είπε. Φαμπρίτσια Λαπικολέλα είναι η πρόεδρος από την Ιταλία. Εντάξει. Ο Πίτερ Γιέτσεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Στα εισαγωγικά σας σχόλια αναφέρατε τις τρέχουσες και μελλοντικές πρωτοβουλίες της Κομισιόν για τη βελτίωση του πλαισίου, του νομικού πλαισίου. Απ' την άλλη πλευρά του νομίσματος όμως έχουμε την εφαρμογή. Κατά την άποψή μου, ένα από τα βασικά προκαταρκτικά ευρήματα αυτής της Επιτροπής είναι ή ενδεχομένως να είναι ότι ο εποπτικός ρόλος της Κομισιόν στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου ήταν κάπως ανεπαρκής ή αμελήθηκε. Ε, μιλάω για το ξέπλυμα χρήματος, τη φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Φαίνεται από τα Panama Papers ότι υπήρχαν σκάνδαλα ε, μεγάλης κλίμακας και δεν είδαμε πολλά από την πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά δηλαδή τη συνεργασία της με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Επίσης φαίνεται ότι η Κομισιόν δεν έχει αρκετές δυνατότητες να αντιμετωπίσει αυτό το εγχείρημα γενικότερα, δηλαδή ε, μία λίστα με τις χώρες υψηλού κινδύνου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πρέπει να βασιστεί η Κομισιόν όχι στον εαυτό της αλλά σε άλλα ε, άλλους θεσμούς. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Όπως ε, ε, καταλαβαίνετε, επειδή δεν έρχεστε συχνά εδώ, ίσως είναι η τελευταία σας ευκαιρία για να μπορέσετε να διασκεδάσετε αυτές τις σοβαρές αμφιβολίες που υφίστανται για το ρόλο της Κομισιόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Έχετε πάλι λιγότερο από τα δύο λεπτά. Έχει δίκιο ο συνάδελφος δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας, είναι και θέμα εφαρμογής. Η νομοθεσία συχνά είναι πιο ισχυρή από την εφαρμογή. Η Κομισιόν όμως σε ό,τι αφορά την οδηγία και τη διοικητική συνεργασία έχει ξεκινήσει 39 διαδικασίες σε παραβάση. Δεν μπορείτε να πείτε λοιπόν ότι ήμασταν παθητικοί και σιωπηλοί. Κάναμε τη δουλειά μας και έχουμε την πρόθεση να παρακολουθήσουμε πολύ στενά την εφαρμογή όλων των οδηγιών που έχουν εγκριθεί από τότε που έχουμε αναλάβει και όλες τις οδηγίες που θα εγκριθούν, ελπίζω, στο μέλλον πριν τελειώσει η θητεία μας. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά σημαντική. Για τη μαύρη λίστα. Ναι, δεν είμαι εδώ για να επικρίνω τα κράτη-μέλη. Έχω συνηθίσει βέβαια να το κάνω, το έχουν συνηθίσει και αυτοί, αλλά εξετάζουμε την δεύτερη εκδοχή τη μαύρη λίστα. Είμαστε σε επαφή με τα κράτη-μέλη. Σκοπεύουμε να τη δημοσιεύσουμε πριν από το τέλο του έτου. Να δημοσιεύσουμε ένα νέο, μια νέα μαύρη λίστα σε ό,τι αφορά τι ε, φορολογικέ ε, φορολογικά συστήματα εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ευθυγραμμίζονται με τα πρότυπά μα. Πολύ ωραία λοιπόν. Πάμε τώρα στους ε, εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Ροζάτη εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και εσάς ε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής που ήρθατε σήμερα εδώ και για την εισαγωγή σας. Δύο γρήγορες και σύντομες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα όμως ε, να επενέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προσπάθειες που κατέβαλε ε, τον τελευταίο 1,5 χρόνο να εισαγάγει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Βέβαια το κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλα αυτά έχω κάποιες αμφιβολίες, θα το πούμε αργότερα.

Στην περίπτωση των Panama Papers διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποια κρατημέλη που ε, σε αυτά εμφανίζονται περισσότερο από άλλα. Κατά την άποψή σας, πού ακριβώς οφείλεται αυτό, οφείλεται ενδεχομένως ε, στο ότι δεν εφαρμόζουν, δεν υιοθετούν την ενωσιακή νομοθεσία ή μήπως αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν κάποια κενά στις δικές τους τις νομοθεσίες που εξηγούν το γεγονός ότι το Λουξεμβούργο ή η Ολλανδία εμφανίζονται πολύ περισσότερο από άλλες χώρες. Ποια είναι η δική σας η άποψη επ' αυτού και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να κλείσει ή δυνατόν αυτά τα κενά. Και η δεύτερη ερώτησή μου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πότε ακριβώς άρχισε να κάνει έρευνες για τα Panama Papers και υπάρχει άραγε μέσα στην Επιτροπή και προς τα έξω παρουσιάστηκε κάποια έκθεση για τα Panama Papers και αν υπάρχει τέτοια έκθεση μήπως θα ήταν δυνατόν να τη διαθέσετε και σε αυτήν την Επιτροπή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφε, ο πρόεδρος Επιτροπής έχει τρία λεπτά στη διάθεσή του για να απαντήσει κατά πόσον έχουμε προβεί σε ενδελεχή ανάλυση όσον αφορά ε, τα Panama Papers, ε, πρέπει να σας πω ότι είμαστε ευχαριστημένοι τουλάχιστον ό,τι έχουμε γράψει ως Επιτροπή δεν έχει διαρρεύσει. Βεβαίως ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν είμαι άμεσα υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Επίτροποι φέρουν την, έχουν την αρμοδιότητα και προτιθέμετα να σας δώσουμε τις απαντήσεις σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω είχατε και μία συνάντηση με τον κύριο Μοσκοπησή. Ε, ε, άντε, θα ξεκινήσω από το χρόνο μηδέν. Λοιπόν, ε, θα πάρετε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που μας κάνετε. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, εμείς όλα τα κράτη-μέλη τα αντιμετωπίζουμε με τους ίδιους όρους, δηλαδή διαδικασίες επί παραβάση. Δρομολογούνται οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο. Και απαντώντας σε αυτό που είπατε, το γιατί κάποια κράτη εμφανίζονται περισσότερο από άλλα στα Panama Papers, θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι γίνεται αναφορά σε διάφορα κράτη-μέλη, ε, αλλά αυτό αναφέρεται στο παρελθόν. Τώρα πια έχει αλλάξει ο κόσμος και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτό που είπατε και αυτό αφορά αυτά τα κράτη-μέλη. Μπας περιπτώσει, θα επανέλθουμε αργότερα επί του θέματος. Προς το παρόν έχουμε καταθέσει 12 νομοθετικές πράξεις, άλλη μία θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες, αλλά θα έχω την ευκαιρία να επανέλθω σε αυτό, γιατί θέλουμε να κλείσουμε τα παραθυράκια, να καλυφθούν τα κενά. αυτό είναι ο στόχος των προτάσεων που έχουμε καταθέσει στο Συμβούλιο. Πολύ ωραία. Επόμενος για τους ε, σοσιαλδημοκράτες ο κύριος Πίτα Ζήμων. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, ε, να αναφερθώ σε αυτά που κάνατε τα τελευταία χρόνια. Εγώ θυμάμαι πάρα πολλές φορές στη Γερμανία, όπου όταν τους έλεγα αυτά που τους έλεγα, οι άνθρωποι δεν με πίστευαν. Ε, γι' αυτό λοιπόν Ας το πούμε ξεκάθαρα. Το όνομά σας ε, συνδέεται με την Ευρώπη με ένα σύστημα, ε, μια χώρα όπου πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδίσει πάρα πολλά χρήματα φορολογικό ντάμπινγκ. Αυτή είναι η εντύπωση που επικρατεί στην Ευρώπη. Και εγώ στη δική μου την εκλογική περιφέρεια, οποτεδήποτε του ενημερώνω ε, το τι έχει κάνει η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια, πραγματικά εκπλήσονται. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάποια ε, στράτευση η οποία ε, αφορά τρεις τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι κατάλογος για τους παραδείσους ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος. Εδώ στην Επιτροπή είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τόσο με τη διοίκηση όσο και με τους αρμόδιους ε, επιτροπές τρόπους ε, για τον κατάλογο αυτό όπου εμφανίζονται χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και το Αφγανιστάν και μια χώρα που δεν έχω ξανακούσει το one wa του κάπως έτσι αλλά εν πάση περιπτώσει όλος ο κόσμος ξέρει ότι αυτή είναι παράδειση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Παναμάς δεν αναφέρεται εκεί και η απάντηση είναι ότι για δύο ολόκληρα χρόνια θα έπρεπε να χρειαστούν πάρα πολλά άτομα για να αξιολογηθεί ε, κατά πόσο θα πρέπει μια χώρα να μπει στον κατάλογο αυτό το να το λέει κανεί αυτό όμω, ξέρετε κάτι, αυτό για μένα σημαίνει ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να εξετάζετε καλύτερα τα πράγματα. Να φτιάξετε μία λίστα, ένα κατάλογο, ε, να αναφέρετε εκεί και ο Πανανάς, να συνεργα... να συνεργαστείτε και με τον Παναμά. Και ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξω αφορά τι φορολογικέ οάσει, ε, ε, του παραδείσου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μήπως μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε να υπάρχει ένα κατάλογο με φορολογικό φορολογικούς παραδείσους ε, όπου θα περιλαμβάνονται και χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπερπόντιων διαμερισμάτων. Τρίτον, ε, ε, επενέσατε τη στράτευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλετε να ζητήσετε από τα κράτη-μέλη να υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις ε, φορολογικές απάτες, γιατί αυτό το χρειάζεστε. Τα κράτη-μέλη βεβαίως ε, δεν το πράττουν αυτό στο βαθμό που η αστυνομία πλέον είναι ο θεματοφύλακας των συνθηκών και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις. Δύο λεπτά ε, χρειαστήκατε. Μήπως μπορείτε να ξαναπαναλάβετε την τρίτη ερώτηση. Δεν την κατάλαβα, λέει ο πρόεδρος Επιτροπής. Πρόκειται για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών η οποία αποφασίστηκε για τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, δηλαδή, ε, τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να ελέγχουν μόνα τους κατά πόσον ε, υπάρχει κάτι που τα επιβαρύνει, γιατί αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη αρνούνται το να υπάρχει ενημέρωση και μεταξύ του ε, και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά η Κομισιόν, ω θεματοφύλακα των συνθηκών, θα πρέπει η Κομισιόν να έχει αυτή τη γνώση για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω με το τρίτο ερώτημα. Γιατί αυτή πραγματικά είναι πολύ σημαντική αυτή η τρίτη ερώτηση. Εμείς είχαμε πει όταν καταθέσαμε την πρόταση για τους φορολογικούς κανόνες, τα tax rulings, ότι η Κομισιόν θα πρέπει να ενημερώνεται για ε, τους υπάρχουν φορολογικούς κανόνες. Αυτό το απέρριψαν κάποια κρατημέλη και εγώ δεν το βρήκα σωστό. Και να σας πω κάτι, θα συνεχίσουμε να, σκύου, να σκούμε πίεση, γιατί πραγματικά χρειαζόμαστε ένα φορέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχει την ε, γενική υποπτία και θα πρέπει ε, οι νομοθετικές ρυθμίσεις να είναι συμπληρωματικές, τροποποιητικές ε, και εγώ επίσης επιθυμώ διακαώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενημερώνεται για τους φορολογικούς κανόνες. Εδώ λοιπόν χρειαζόμαστε απαραίτητα τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη όπως επίσης και με άλλους άμεσα θυγόμενους. Γιατί όποιος ανακοινώνει κάτι στην εφορία του, στη φορολογική του αρχή, αυτό ε, να το ανακοινώνει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να το κάνει ο ίδιος, να το πράττει η φορολογική αρχή της χώρας. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι, και νομίζω ότι το έχω πει αυτό, πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε μια συμπλήρωση και ολοκλήρωση του καταλόγου των φορολογικών παραδείσων. Πρέπει να ολοκληρωθεί λοιπόν αυτός ο κατάλογος με τους φορολογικούς παραδείσους. Αλλά επιτρέψτε μου να επισημάνω κάτι. Το είπα αυτό, το είπα στα γερμανικά, λέει ο κύριος Γιούνκερ. Δεν το είπα στα γαλλικά, στα γερμανικά το είπα. Τώρα όμως θα συνεχίσω στα γαλλικά. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχουμε τους ανθρώπινους πόρους πραγματικά για να προβούμε σε τέτοιου είδους εξέταση. σε σχέση με κάποιες κοινωτικές ομάδες δεν έχω τόσο εξοπλισμό, τόσα μέσα, οπότε δεν μπορώ να σας ε, υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν μπορώ να τηρήσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να επιληφθεί του θέματος ε, για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Και κατά τα άλλα να σας πω ότι εμείς εξαρτώμεθα και από την καλή βούληση των κρατών μελών. Γιατί κάποια κρατημέλη έχουν πληροφορίες για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τρίτες χώρες και θα ήταν χρήσιμο να ανακοινώσουν τις πληροφορίες αυτές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν ε, να γνωρίζουμε την άποψη των κρατών μελών, ποιοι είναι η φορολογική παράδοση, ακόμα και αν δεν συμφωνούν όλοι επί του καταλόγου των φορολογικών ε, παραδείσων. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τρίτες χώρες ε, οι οποίες ε, είναι υπέτειες για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Πολύ ωραία. Επόμενος στον κατάλογό μου, ο κύριος Μπέρντ Λούκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Γιούνκερ. Είπατε στις εισαγωγικά σας ε, σχόλια ότι από τα Panama Leaks ε, ξέρετε σε ποιο μέγεθος υπάρχει φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή από τις πολυεθνικές. Να πω ότι ε, πολλοί από εμά το ξέραμε από πριν. Ήταν ένα ανοιχτό μυστικό ότι ε, όποιος ήθελε να σώσει χρήματα από την εφορία πήγαινε στο Λουξεμβούργο. Εσείς μέσα από τα Panama Leaks όμως το μάθατε ότι υπήρχε αυτή η τεχνική της ε, φοροδιαφυγής, ενώ εμείς το ξέραμε από πριν. Το ξέρατε λοιπόν από πριν, από το 2003, τότε που είχαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις καταθέσεις, ε, γνωρίζατε ήδη το πρόβλημα. Όταν το μάθατε λοιπόν, γιατί δεν έκανε το Λουξεμβούργο την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με την οδηγία, γιατί ε, καταλαβαίνετε ότι πέρα από το Λουξεμβούργο υπήρχαν και άλλες χώρες που ασκούσαν αυτή την ε, πολιτική. Αυτό έκανε το Λουξεμβούργο, άρα μπορούσαν και οι υπόλοιπε. Δεύτερα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το Panama Leaks, αλλά και με το Luxembourg Leaks ε, για τα tax rulings ε, μέσα, σε, μέσα από τον εργαλείο του ανταγωνισμού μπορέσαμε να έχουμε διαστρέβλωση του ανταγωνισμού στο ευρωπαϊκό επίπεδο και η Κομισιόν δεν χρησιμοποίησε τα εργαλεία που είχε για να μπορέσει να εξετάσει αυτό το θέμα. Υπήρχε πάντοτε μια ε, επιλεκτική στάση. Σε κάποιες περιπτώσεις δηλαδή ε, επεξεργαζόταν το θέμα, σε άλλες όχι. Αν ξανασκεφτούμε λοιπόν αυτό το θέμα, αυτές οι tax rulings ε, θα αν το είχαν ασκηθεί σωστά οι διαδικασίες θα μπορούσαμε να είχαμε ε, προλάβει αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά. Κοιτάξτε, υποβάλλατε πάρα πολλές ερωτήσεις, ε, αλλά θα επανέλθω καταρχήν σε αυτά που είπε ο κύριο Σίμων, γιατί μου έθεσε το ερώτημα κατά πόσον ε, και ε, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν φορολογική παράδοση, παράδειση και κατά πόσο θα πρέπει να τους αποκαλύψουμε όχι. Όχι, δεν θα τους αποκαλύψουμε. Γιατί, ξέρετε κάτι, αυτό σας λέω αφορά το παρελθόν, δεν αφορά το μέλλον. Ως εκ τούτου εμείς δεν θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε αυτό, εκτός αν προκύψουν αποχρόντες λόγοι και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ονοματίσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τώρα, να σας εξηγήσω για δύο λεπτά, μέσα σε δύο λεπτά, ε, γιατί το Λουξεμβούργο ακολούθησε ένα διαφορετικό φορολογικό μοντέλο από ό,τι άλλες χώρες ε, και γιατί εξακολουθεί να ισχύει το τραπεζικό απόρριτο, δεν μπορώ να το κάνω σε δύο λεπτά. Αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι παλαιότερα ζούσαμε σε ένα διαφορετικό κόσμο και τότε παρεπιπτόντως και η επιστήμη στην, στους επιστημονικούς κύκλους ε, επικρατούσε η άποψη ότι το να υπάρχει παρακράτηση φόρου στην πηγή, κατ' ουσίαν αυτό σημαίνει κατάργηση του τραπεζικού απόρριτου. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο το να επιβληθεί φόρου στην πηγή του ύψους του 35% αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο κάτω από ορισμένε συνθήκες και μόνο αν οι χώρες Μπενελούξ θα μπορούσαν να περάσουν σε ένα σύστημα που οι ίδιες χώρες θα καθόριζαν. Και οι προποθέσει αυτέ ξέρετε ποιες ήταν. Δηλαδή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε υποχρεωμένοι να φορολογούμε τα κέρδη που προκύπτουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σύστημα αυτό δεν αφορά μόνο τις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τρίτες χώρες, Αντόρα, Σαν Μαρίνο και ού αυτό αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα έπρεπε να εμπλακούν σε αυτό το σύστημα της αυτόμητης ανταλλαγής πληροφοριών. Αν βέβαια είχαν ισχύσει όλα αυτά τότε το 2002 πράγματι θα μπορούσε να υπάρξει συνύπαρξη δύο διαφορετικών συστημάτων. Παρεμπιπτόν να πω κιόλα ότι τότε είχε συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. Εντάξει δεν ήταν ε, ε, η διαδικασία του συναπόφαση. τότε όμω είχε ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Κοινοβούλιο είχε συνενέσει και είχε πει ναι εντάξει να υπάρχουν αυτά τα δύο παράλληλα συστήματα. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι αρμόδιο για θέματα ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Όταν όρισα αρμόδια επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού,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 τη είπα ότι ποτέ, μα ποτέ, και το έχω τηρήσει, ποτέ δεν θα ανθίξω θέμα ανταγωνισμού. Και ήξερα πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ερευνούσε για κάποιες περιπτώσεις που αφορούν το Λουξεμβούργο. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ήθελα ούτε στο παραμικρό να δώσω την εντύπωση ότι πραγματικά προσπαθώ να προστατεύσω το Λουξεμβούργο. Γι' αυτό η κυρία Μπεστάγκερ είναι απόλυτα ανεξάρτητη. Βεβαίως και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους επιτρόπους ανθρώπου και είναι πάρα πολύ καλή στη δουλειά τη. Τώρα, γιατί ορισμένε περιπτώσει εξετάζονται πιο αυστηρά από άλλε, ε, απευθυνθείτε στην ε, κυρία Επίτροπο. Μην με ρωτάτε εμένα για αυτά τα θέματα. Δυστυχώς ετέθη μια ερώτηση εκτός μικροφώνου. Η απάντηση του κυρίου Πρόεδρου είναι ότι μίλησα για δυνατότητα ανασύνθεσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν μου ανακοινωθεί ότι δεν επαρκούν οι πόροι της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας, ε, παρότι ε, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό έχει αποδειχθεί, τότε προφανώς θα υπάρξει η αναδιάρθρωση και η ανασύνθεση. Αυτά που είπατε ε, σχετικά με τις αποταμιεύσεις το ήξερα αυτό. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο προσπαθήσαμε να λύσουμε το θέμα ήδη από το 99. Εγώ ήμουν τότε πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ και είχα πει ότι οι αποταμιεύσει θα πρέπει να φορολογούνται στο σύνολο της, ε, των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν ήξερα το πώς οι Γερμανοί θα μεταφέρουν τα λεφτά του στο Λουξεμβούργο, ούτε και πώς οι Λουξεμβούργοι είχαν επενδύσει στη Γερμανία. Οι αποταμιεύσει θα πρέπει να φορολογούνται παντού με τον ίδιο τρόπο. Αλλά τότε παλαιότερα, αν θυμάστε, ε, οι μη υπήκοοι μιας χώρας δεν φορολογούνται τουλάχιστον ως προς τις αποταμιεύσεις τους. Επόμενος στον ε, καταλογό μου εκ μέρους των φιλευταίων είναι ο κύριος ε, Τόιρεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Θα σας πω τελείως ειλικρινά. Αυτά που μας είπατε αρχικά με απογοήτευσαν απογοητεύτηκα. Κατά την άποψή μου χάσαμε μία ευκαιρία και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μία ξεκάθαρη ερώτηση. Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες και ενδιαφέρει και εμάς είναι το εξή. Οι αποκαλύψεις του, των Panama Papers τι έδειξαν. Έδειξαν ότι έχουμε συγγενείς ε, του Πούτιν, του Ασάντ, φίλοι τους, ε, οι οποίοι βρίσκονται σε κάποιους καταλόγους ε, δίωξη. Πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, πρόκειται για εικονικές εταιρείε. Το θέμα λοιπόν που τίθεται είναι Ποιο αναλάβει την ευθύνη, τη δικαστική αλλά και την πολιτική ευθύνη. Και στα Panama Papers αναφέρεται ότι μια χώρα που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, δηλαδή το Λουξεμβούργο, βρίσκεται σε τέταρτη θέση όσον αφορά τους διαμεσολαβητές. Είναι πάνω από 15.000 οι διαμεσολαβητές του Λουξεμβούργου, μεταξύ αυτών και η Μονσάκ Φωσέκα. Ερωτώ λοιπόν ξεκάθαρα, ποιος φέρει την πολιτική ευθύνη. Και ε, Πώς θα το επεξεργαστούμε αυτό. Ε, τα βρίσκεται όλα ικανοποιητικά. Αν είναι σωστά να μην τα ερευνήσουμε. Αλλά η Επιτροπή με εσά που είσαστε πρόεδρος της, τι ακριβώς θα κάνει για να αποκαλυφθούν στοιχεία. Πρόεδρος, επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι. Όταν εμείς πήγαμε στο Λουξεμβούργο, τότε ο δικηγορικός σύλλογος μας είπε ότι αυτοί που είναι στα Panama Papers και δεν είναι τράπεζες, δεν είναι 14.000 τα ονόματα, είναι 2.500. Κύριε Τζούγκερ, σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Δεν τα ξέρω αυτά που είπατε και είπα προηγουμένω ότι έχουμε αναλάβει 12 νομοθετικέ πράξει Τον Ιούνιο θα καταθέσουμε άλλη μία και αυτή ακριβώ αφορά του intermediaries, του διαμεσολαβητές ε, που αναφέρετε προηγουμένω. και αυτοί σχετίζονται όχι με το Λουξεμβούργο αλλά και κοντά στο Λουξεμβούργο υπάρχουν και άλλοι πολλοί intermediaries που ασχολούνται με τέτοια θέματα. Πρέπει λοιπόν να του αντιμετωπίσουμε και αυτό θα το με πρόταση οδηγίας που θα κατατεθεί τον Ιούνιο. Και επιθυμούμε το αργότερο, την 1η Ιανουαρίου του 2019, να τεθεί σε ισχύ αυτή η οδηγία. Γιατί πραγματικά είναι πρόβλημα και δεν είναι δυνατόν να κρύβεται κανείς πάντα πίσω από το απόρριτο, το δικηγορικό όταν θέλει να επεξεργαστεί τέτοιου είδους προτάσεις ο κύριο Τόρερ θα κάνει μια συμπληρωματική ερώτηση. Αλλά εσεί τι θα πείτε στου πολίτε, την πολιτική ευθύνη, Ποιο τη φέρει, Ποιο δεν την αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Κύριε Γιούγκερ, εγώ δεν νομίζω ότι στον ε, πολιτικό τομέα θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνε. Διότι, όπως λέμε και στα γαλλικά, οι, πολιτικά, πολιτικοί ηθήνοντες ε, δεν ε, είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να παρέμβουν στο θέμα των διαμεσολαβητών. Ο Πρωθυπουργό ε, του Λουξεμβούργου και οι Υπουργοί δεν έχουν στα χέρια τους εμπορικό μητρό, δεν το κρατάνε αυτοί. Τώρα, με την αποκάλυψη βέβαια μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα δρόμους και παρακάμψεις στις οποίες κινούνται οι ε, intermediaries και θα πράξουμε τα δέοντα. Επόμενος ομιλητής για την ΚΟΕΑ Φάμπερ Ντιμάζες. Η τελευταία συνάντησή μας, ε, ε, αν θυμάμαι καλά, επισκιάστηκε από αυτές τις εκθέσεις Κρέκερ για τις ε, tax rulings στο Λουξεμβούργο. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ στο μέλλον. Είπατε ως πρόεδρος της Κομισιόν επειδή δεν έχουμε κάθε φορά την ε, ευκαιρία να σας ε, μιλάμε ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως πρώην Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορέσετε να μας δώσετε τα έγγραφα από τις ομάδες Code of Contact, αν μας λέτε ότι δεν υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι στην Ευρώπη, να μας τα δείξετε για να μην μας τα κρύβετε. Επίσης, η οδηγία για τους τόκους και πάλι ήταν εξαίρεση το Λουξεμβούργο και ε, ως ε, ε κάτοικοι της Ευρώπης μπορεί κανείς να έχει έναν λογαριασμό νομική, νομικό πρόσωπο στο Λουξεμβούργο. Τι έχετε να πείτε και για αυτή την εξαίρεση. Επίσης είπατε στη Φορολογική Επιτροπή στο παρελθόν ότι δεν ε, συζητάμε φορολογικές υποθέσεις. Ε, ποτέ δεν έγινε αυτό, όμως από το Internal Revenue Service ε, το Σεπτέμβριο του 2013 είχατε μιλήσει με την Amazon και είχατε χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό συζητώντας για το Λουξεμβούργο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι είπατε σε αυτή τη συζάτηση για τη φορολογική πολιτική θέματα του Λουξεμβούργου. Ο Υπουργό Οικονομικών της Μαδέρα μα είπε ότι το 2010 η πρεσβεία του Λουξεμβούργου είχε πάει στη Μαδέρα με μια λίστα από εταιρείε ε, που είχαν 5% φορολογία και θέλαν να πάνε στην, ε, από τη Μαδέρα στο Λουξεμβούργο. Ο πρέσβης του Λουξεμβούργου ε, το έκανε αυτό από μόνος του ή ήταν μια επιταγή της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου. Ήταν απλώς ένας διπλωμάτης που το έκανε αυτό. Μας είχατε πει πώς περάσαν όλες αυτές οι πληροφορίες με email, με Learjet, προσωπικά. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, αυτά που είπατε σήμερα αποδεικνύουν ότι έχετε κάποια κενά μνήμης. Εγώ όμως δεν θα σας τα υπενθυμίσω. Εγώ ε, το μόνο που θέλω να πω ότι δεν έχω καταγράψει σε χαρτί πότε ο κύριος Κρέκε μου έδωσε αυτό χαρτί σε, ποια, σε ποιο σημείο, σε ποιο μέρος, τι ώρα. Αν όμως ε, τον συναντήσω θα του πω να μου, θα του ζητήσω να μου πω ε, πώς ακριβώς απέκτησε αυτό το χαρτί. Τέλος πάντων, σημασία τι έχει τώρα, ότι υπάρχει αυτό το χαρτί και όχι πώς έφτασε σε μένα. Ε, νομίζω ότι δεν έχει νόημα τώρα να μπούμε στη λεπτομέρεια πώς ακριβώς έφτασε αυτό το χαρτί στα χέρια μου. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι δεν έχω μιλήσει με κανέναν για φορολογική φύσεω θέματα. Άλλο είπα. Είπα ότι εγώ ποτέ δεν πλάκιν στην φορολογία μιας εταιρεία. Όταν, αν πάτε στο εξωτερικό, θα σας ε, τεθούν τέτοιου είδους ερωτήσεις. Πολύ θα μας άρεσε ε, να έρθει η Amazon στο Λουξεμβούργο. Δεν το αμφισβητώ αυτό, αλλά όχι ότι εγώ ήρθα σε επαφή με την Amazon, γιατί αυτό δεν είναι δουλειά του Υπουργού Οικονομικών που ήμουνα τότε. Δεν ήμουνα ο αρμόδιος, γι' αυτό λοιπόν εγώ απάντησα σε ερωτήσεις, αλλά σας λέω ποτέ μα ποτέ εγώ δεν έλαβα συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα για μία εταιρεία στο Λουξεμβούργο υπάρχει ένας άκαμπτος κανόνας. Αρμόδιες είναι οι φορολογικές αρχές για θέματα ε, φορολόγησης και όχι ο υπουργό Οικονομικών. Τώρα, όσον αφορά τα tax rulings στο ε, Λουξεμβούργο, σας είπα, ε, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι. Σε άλλες χώρες είναι αρμόδιοι Υπουργό Οικονομικών. Πριν με ρωτήσετε, να μαθαίνατε, αλλά εντάξει, Κύριε Πρόεδρε, ε, λυπάμαι, ο πρέσβης όμως του Λουξεμβούργου, γιατί γι' αυτόν εγώ σας ρώτησα, που πήγε στην Πορτογαλία, αυτό δεν είναι φορολογική αρχή. Κοιτάξτε, οι διπλωμάτες ε, πάγονται στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και δεν μπορώ να φανταστώ τώρα ότι ο κύριος Άσελμπον, ο Υπουργός Εξωτερικών, έδωσε εντολή στον πρέσβη να πάει στη Μαδέρα και να αρχίσει να κάνει τον γύρο των εταιριών. Κάτι διάβασα κι εγώ, ε, πράγματι ε, στο Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου έχει κατατεθεί επερώτηση για τον Υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου που δεν είναι στο Λουξεμβούργο, κάπου αλλού είναι. Όταν επιστρέψει θα απαντήσει σε αυτή την προφορική επιρώτηση. Εν πάση περιπτώσει είναι θέμα της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου να απαντήσει. Το ότι Πήγα το Δεκέμβρη του 2003 εγώ στην Ουάσιγκτον. Πρώτη φορά τα ακούω. Επόμενος για τους πράσινους ο κύριος Σβέν Κίγκολτ. Κύριε Πρόεδρε της ε, Επιτροπής, ε, είδαμε πολύ προσεκτικά το τι ακριβώς ε, αναφέρεται για την φορολογία ιδιωτών στο Λουξεμβούργο. Τι έγινε ακριβώς τα τελευταία χρόνια. Και διαπιστώσαμε ότι η οδηγία περί επιτοκίων που ήταν αντικείμενο σκληρών διαπραγματεύσεων στο Κοινοβούλιο και παρεπιπτόντος με την επιθυμία του Λουξεμβούργου να υπάρχει ένας φόρος της τάξης του 10%. Τέλος πάντων λοιπόν αυτή η συγκεκριμένη οδηγία όμως παραβιάζεται. Και με βάση τα στοιχεία τα οποία αναλύσαμε ο κύριος Λάγκεν συμμετείχε, διαπιστώσαμε ότι οι παραβιάσεις λαμβάνουν χώρα κυρίως στο Λουξεμβούργο και όχι στο Βέλγιο ή στην Αυστρία. Αυτή η παράκαμψη μέσα από ε, ασφαλιστικές εταιρείες και μέσα από υπεράκτιες ε, εταιρείες, όλα αυτά οδήγησαν στο να προχωρήσει ακόμα πιο πέρα η φοροδιαφυγή και η αποφυγή. ερωτώ λοιπόν το εξής κύριε Γιούγκερ, εσείς στα κράτη-μέλη τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους φοροφυγάδες και στο Λουξεμβούργο και αλλού. Θα τις βοηθήσετε τις χώρες αυτές έτσι ώστε στο πλαίσιο της διοικητική αρρωγής να καταστεί δυνατόν αυτούς τους διασυνοριακούς φοροφυγάδες, οι χώρες που ενδιαφέρονται να τους εντοπίζουν και μετά να ακολουθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Και δεύτερη ερώτηση. Μετά τα Panama Papers στη Γενική Διεύθυνση Δικαίου έχουμε μια task force που ασχολείται με την χρηματοψηφιακή εγκληματικότητα και εκεί απασχολούνται έξι άτομα. Σήμερα υποσχεθήκατε να αυξήσετε το προσωπικό αυτή τη task force για να κάνουν καλή δουλειά. Και τελευταία ερώτηση κράτη-μέλη, υπάρχουν κράτη-μέλη ε, που δεν εφαρμόζουν κάποιες προτάσεις που καταθέσατε. Εσείς λοιπόν, σας ερωτώ, αυτά που μπλοκάρουν ε, τα κράτη-μέλη, είσαστε πρόθυμος να εφαρμόσετε το άρθρο 116, είσαστε πρόθυμος ε, να περάσετε στην διαδικασία την πλειοψηφική, γιατί σε τελική ανάλυση μια τέτοια απόφαση της Κομισιόν θα οδηγήσει στο ορισμένα κράτη-μέλη να δηλώσουν τη θέση τους και να μην κρύβονται πίσω από φορολογικούς παραδείσους. Η απάντησή μου είναι πολύ απλή και στις τρεις ερωτήσεις σας ναι, ναι, ναι και πάλι ναι. Τρία ναι. Πολύ ωραία, ξεκάθαρη η απάντηση. Ναι σε όλα λοιπόν. Ο κύριος Γκέγκολτ όμως θα ρωτήσει συμπληρωματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μας είπατε. Εμείς θα συνεχίσουμε τις έρευνές μας. Να σας πω όμως κάτι. Αυτό που επιθυμούν ε, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι αυτό που μόλις τώρα είπε ο κύριος Τόιρ. Θα το πω ξεκάθαρα. Εσείς ε, πάτε από τον Άννα στον Καϊάφα και το δουλεύετε αυτό. Μέχρι σήμερα όμως οι πολίτες θέλουν να αναλάβετε την ευθύνη. Και Κατ' ουσίαν, αυτό είναι αυτό που σας επιβαρύνει. Επιβαρύνει την αξιοπιστία σας. Και το λυπάμαι, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί εντωμεταξύ πρέπει να ομολογήσω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση, προς την φορολογική συνεργασία. Συνάδελφε Γκίγκολτ, έχω κάθε κατανόηση για το ότι επιθυμείτε να αναφερθείτε και στο παρελθόν σε αυτό το θέμα, που είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα ήθελα όμως την αξιοπιστία μου να την κρίνετε εσείς ε, με βάση τη λάσπη που διασπείρετε έναντί μου την αξιοπιστία μου και αυτή τη Επιτροπή θα πρέπει να την κρίνεται με αυτά που πράττει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι καμία άλλη επιτροπή δεν έχει αναλάβει τόσε πολλέ πρωτοβουλίε για τη φοροαποφυγή. 12 είναι. Αν θέλετε και να σα τι απαριθμίσω για να μην τι ξεχνάτε. Λοιπόν, το Μάιο του 2015 είχαμε μία νέα οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τα tax rulings. Αυτή η οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2017 και από το Σεπτέμβριο του 2017 θα έχουμε την, την πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κατόπιν τον Ιανουάριο του 2016 καταθέσαμε προτάσεις για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με βάση τις ε, country by country reports, ε, εκθέσεις των πολυεθνικών ελληνικών Μια τέτοια πρόταση δεν είχε γίνει ποτέ. Επίσης ε, προτείναμε και Νομίζω αυτό δεν χαροποίησε πολλούς, αυτές οι country by country reports να δημοσιοποιούνται. Αυτή την πρόταση την καταθέσαμε τον Απρίλιο του 2016 και ευτυχώς το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2017, δηλαδή 7-8 μήνες αργότερα, ε, στην αρμόδια επιτροπή επιλήφθηκε του θέματος κάτι ε, το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερα. Αργότερα, τον Ιούνιο του 2016, καταθέσαμε περαιτέρω προτάσεις για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και τον Ιούλιο, τον ίδιο μήνα δηλαδή του 2016, θεσπίσαμε νέους ε, κανόνες για fiscal information, για την ε, κατάθεση πληροφοριών στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Αργότερα, θεσπίσαμε ένα νέο πλαίσιο για τη διαφάνεια με την ε, Ελβετία, το Σαν Μαρίνο, την Ονδούρα. Αυτά έγιναν είχαν, ακολούθησαν αφού είχαν ήδη προηγηθεί πάρα πολλές άλλες ε, πρωτοβουλίες. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2016 θεσπίσαμε την οδηγία Anti-Tax Avoidance, την ενισχύσαμε περισσότερο την οδηγία αυτή και τον Οκτώβριο του 2016 καταθέσαμε και άλλες ε, συναφείς προτάσεις. Εξάλλου, καταθέσαμε νέες προτάσεις για την φορολογική βάση και Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει συνέχιση του θέματος αυτού. Κατόπιν τον Οκτώβριο του 2016 ασχοληθήκαμε με την αποφυγή της διπλής ε, φορολογίας και τον, ε, το 2019 αυτή η, ε, αυτός ο μηχανισμός διευθέτησης διαφορών θα τεθεί σε ισχύ. Κατόπιν, επίσης, τον Ιανουάριο του 2016 καταθέσαμε ένα κατάλογο για non-cooperative tax tax jurisdictions. Αυτός ο κατάλογος πρέπει να συμπληρωθεί. Αυτό θα γίνει πριν από το τέλος του έτους και τον Ιούνιο αυτού του έτους θα καταθέσουμε άλλες ε, προτάσεις για αφρολογικά θέματα. 13 λοιπόν οι πρωτοβουλίες τις οποίες η Κομισιόν ανέλαβε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόεδρος, νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε ότι πράγματι η Κομισιόν προχώρησε. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και εμείς το στηρίζουμε αυτό. Επ' αυτού δεν υπάρχει καμία φιβολία. David Coburn, εκ μέρους της πολιτικής ομάδας EFDD. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά που είστε εδώ κύριε Γιούγκερ. Ως Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου φαίνεται ότι πιστεύατε με μεγάλο ενθουσιασμό στην φορολογικό ανταγωνισμό. Πολύ καλά. Συμφωνώ μαζί σας για την ε, αποδοτικότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρότερα ώστε να είμαστε αποδοτικοί στο να βρούμε τα χρήματα είτε των ιδιωτών είτε των εταιριών και να τα φορολογήσουμε. Τώρα, ως Πρόεδρος ε, της Κομισιόν, έχετε αλλάξει την στάση σας και δεν ασχολείστε με τον ανταγωνισμό. Είστε ο νέος Ζαν ε, Κλοντ. Όπως είπε και ο κύριος ε, Γκίγκολτ, ε, ε, ε, εσείς ήσασταν ένας από αυτούς που άλλαξε τη στάση του ε, έτσι ξαφνικά. Γιατί έγινε αυτό. Θα ήθελα να επανέλθουμε στον παλιό καλό Jean-Claude Juncker που είχαμε τη ανταγωνισμό στην Ευρώπη και την αποτελεσματικότητα που έχει η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε για την ερώτηση. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. David, πραγματικά αναρωτιόμουν πότε θα επανέλθει στη Βρετανία και είδα ότι το έκανε στο τέλος δεν με απογοήτευσες. Όταν με περιγράφεις ως έναν σχιζοφρενή ο οποίος άλλαξε από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν ξέρω, πιστεύω στον φορολογικό ανταγωνισμό που είναι και μία από τις αρχές ε, της συνθήκης. Συνεχίζω. Όμως ε, μαζί με κάποιους άλλους. Ε, δεν θέλω απλώς να αμελήσω αυτή τη διάσταση, απλώς επικεντρώνουμε στον δίκαιο φορολογικό ανταγωνισμό που πρέπει να είναι δίκαιος. Δεν ήταν πάντοτε και δεν ήταν γιατί είχαμε κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, την ε, οδηγία PAT. Εγώ ήμουν αυτός που το 1991 στην ουσία οδήγησα το ECOFIN να αποφασίσει αυτή την οδηγία. Είχαμε 250 διαφορετικά εργαλεία στις διάφορες χώρες για το VAT, για τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Όταν μιλάμε λοιπόν για εξαιρέσεις ε, στις ε, αρχές, ε, δεν νομίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του παλιού και του νέου Γιούγκερ. Απλώς εγώ επικεντρώνομαι στην δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Για το ΙΕΝΕΦ, e Μάριο Μπογκέτσιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πολλές ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και στο χρηματιστήριο γίνονται κρύβοντας ε, τις ε, πραγματικές εταιρείες ε, και την ε, πραγματική προέλευση των χρημάτων. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι πώς, τι ακριβώς μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι στα κράτη-μέλη και κυρίως στους φορολογικούς παραδείσους όπως είναι το Λουξεμβούργο δεν θα συγκεντρωθούν τραπεζικές συναλλαγές χωρίς να ελέγχεται η προέλευση των κεφαλαίων. Και ξέρετε, ε, σαφώς ε, όλα αυτά δεν θα πρέπει να τα δει κανεί μόνο κάτω από το πρίσμα της ε, φοροαποφυγής αλλά και κάτω από το πρίσμα του να παρισφρίουν στην πραγματική οικονομία εγκληματικά κεφάλαια. Και κάτι άλλο. Προκύπτει από αυτό το το κουτί της Πανδώρας που άνοιξε με, τα, με το σκάνδαλο Panama Papers. Μία εταιρεία υποτίθεται ανήκει στο Μουσκάτ, Μουλιέρ, ε, σύζυγο του Πρωθυπουργού. Όμως, ε, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μία εξωχώρια στο Ντουμπάι και εκείνης και της ε, κόρης του δικτάτορα του Αζερβαϊτζάν. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία γιατί ο νέος Γιούνκερ είναι ένας πολεμιστής που έχει βγάλει το σπαθί του για να λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πώς θα χρησιμοποιήσετε το σπαθί σας έχοντας κατά νου όλες αυτές τις πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι περιπτώσεις ε, της κυβέρνησης Μάλτας συζητήθηκαν, αλλά παρακαλώ. Κοιτάξτε αγαπητέ συνάδελφοι, εγώ δεν μπορώ να σα πω ε, όλα αυτά που αφορούν στη Μάλτα. Αυτά δεν αφορούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφορούν, αφορούν τις αρχές της Μάλτας. Αυτοί να επιληφθούν του θέματο. Τα έχω ακούσει και εγώ αυτά, αλλά τώρα τι να κάνω. Έτσι ξαφνικά εγώ να τοποθετηθώ σε κάποιε διαδικασίε που εσεί αναφέρετε στην περίπτωση που ισχύουν. Α πάω τώρα στα άλλα. Όσον αφορά τις πληροφορίες για τους ε, ωφελούμενους, για τους δικαιούχους. Τον Ιούλιο του 2016 προτείναμε νέους κανόνες για να μπορέσουμε να επεκτείνουμε την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στις πληροφορίες για τους δικαιούχους, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό οι φορολογικές αρχές να μπορούν να βρουν ποιος είναι ο τελικός ε, ιδιοκτήτης ε, μιας, ε, ενός προσώπου, μιας νομικής οντότητας. Το 2018 θα μπουν σε εφαρμογή αυτά. Μια επερώτηση ενδεχομένως. Θα κάνω μόνο ένα σχόλιο. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι ο πρόεδρος παραδέχεται ότι αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι μαφίες και οι διάφορες εγκληματικές οργανώσεις μπορούν να επενδύσουν μέχρι το τέλος του 2018 στην πραγματική οικονομία χωρίς κανένα πρόβλημα γιατί κανείς δεν θα τους ελέγχει και δεν έχει και καν την αρμοδιότητα να τους ελέγχει. Αυτό είναι την πρόταση, την κάναμε τον Ιούλιο του 2016 πρέπει να μεταφραστεί στις εθνικές νομοθεσίες η οδηγία. Χρειάζεται μια περίοδος, 1,5 χρόνος, ο οποίος ε, θα ε, είναι στο ενδιάμεσο, παρόλο που είναι το θέμα επίγον. Ευχαριστώ κύριο Φέμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Ε, θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπατε, ότι εκπροσωπώ μια περιοχή όπου το Λουξεμβούργο είναι πολύ μακριά, ξέρετε όμως ποια είναι κοντά, η Αυστρία. Η Αυστρία και τα λεφτά πήγαιναν παλαιότερα στην Αυστρία και στην Ελβετία και όχι στο Λουξεμβούργο. Ε, δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο, υπάρχουν πολλοί αμαρτωλοί στον κόσμο αυτό. Να πω κάτι άλλο όμως, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα φορολογικό παράδεισο και αυτός είναι η Μαντέρα. Συγκεκριμένα στις 27 Μαΐου του 87 για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδέχτηκε το φορολογικό καθεστώς της Μαντέρα. Έγραψε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η άδεια αυτή δεν σημαίνει που δεν είναι ότι συνενεί η Κομισιόν στο να υπάρχει ένας χώρος ε, και μια μια περιοχή για την εγκατάσταση υπεράκτιων εταιριών. Κατ' ουσίαν, περί πρόκειται, πρόκειται για το ότι θα έπρεπε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Το 2014 όμως ε, είχαμε 1.866 εταιρείε ε, και 22.000 θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν. Δηλαδή, ε, πρόκειται για διευθυντές, για υψηλά στελέχη οι οποίοι ε, διαχειρίζονται πάνω από 100 εταιρείε. Και ο Υπουργό Οικονομικών της Μαδέιρα μας είπε ότι στη Φουνχάλ ε, σε ένα συγκρότημα Εκεί έχουν εγκατασταθεί 180 εταιρείε. Το ερώτημα λοιπόν που με απασχολεί είναι ποια μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε αυτά που είπε στο πρώτο έγγραφο έγκρισης το 87 ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν για να υπάρχουν θέσει απασχόλησης και όχι για να εγκατασταθούν εταιρείε υπεράκτης. Τι έκανε η Κομισιόν, το έλεγξε, συμφωνεί με αυτά τα οποία εντωμεταξύ έχουν προκύψει κύριος Γιούγκερ. Αγαπητέ Μάρκους, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πια να ανησυχείς ε, για το θέμα αυτό. Το Klein Weisertal είναι μια περιοχή από εκεί έρθει και γι' αυτό δεν θα πρέπει να ανησυχήσει, γιατί εκεί δεν χρειάζεται να καταβάλουν οι διερχόμενοι διόδια. Ας τα αφήσουμε αυτό. Πάμε στο θέμα. Ε, ο κύριος Ντελόρ ήταν νομίζω αρμόδιος τότε που έκανε αυτή την ε, έγκριση που έδωσε την άδεια. Και τότε ισχύει και ισχύει όμως ακόμα και τώρα ότι για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές χρειαζόμαστε κάποιες ειδικέ ρυθμίσεις. Αυτό ίσχυσε τότε για τη Μαδέρα, ισχύει και τώρα βέβαια. Ε, θυμάμαι Έχω καλή μνήμη, αλλά δεν μπορώ έτσι ξαφνικά να αιτιολογήσω όλες τις αποφάσεις Κομισιόν και πριν από την ε, πτώση του τείχους ε, το 89, εντάξει θα ενημερωθώ. Τι να πω τώρα ας πούμε. Στην ε, Μαντέιρα αυτός που όμως στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθείτε θα είναι στον Υπουργό της Οικονομικών και όχι στην Κομισιόν. Ε, κοιτάξτε, αυτή η άδεια είχε και κάποιο χρονικό ε, περιορισμό, ανανεωνόταν όμως συνέχεια και με τον κύριο Μπαρόζο. Υπάρχει και ένα μνημόνιο συναντήληψης που συνήθει, όπου αναφέρεται και εκεί συμμετείχε και η Τρόικα ότι θα πρέπει να την χάνουν ε, εξέτασης και σε τα φορολογικά καθεστώτα. Άρα δηλαδή το συζητήσατε. Το συζητήσατε και στην Επιτροπή και στο Eurogroup. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από ό,τι μας λέτε. Και δεύτερον, η Κομισιόν οποτεδήποτε χορηγεί μια τέτοια άδεια οφείλει να μεριμνά έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην άδεια. Θα επανέλθω στο θέμα της ε, Μαδέιρα και παρότι τότε συμμετείχα στο Eurogroup δεν ήξερα ότι στις αποφάσεις της ε, Τρόικα για την ε, Πορτογαλία υπάρχει και κάτι για την Μαδέρα. Γιατί αν τοποθετήθηκε η Τρόικα τότε, μάλλον έκανε και κάτι το σωστό. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Τώρα, κλείσαμε με τις πολιτικές ομάδες. Τέσσερις ε, έχουμε catch the eye. Κανονικά για το catch the eye ε, δίνουμε ένα λεπτό. Ξεκινώ με τον Λουί Μισελ. Ναι κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τις διευκρινήσεις που μας δώσατε. Εγώ θα ήθελα πάντως να το δώσω στην εξή μαρτυρία. Η Επιτροπή σας έκανε πολλά περισσότερα από, σε σχέση με άλλες επιτροπές για το θέμα το οποίο εξετάζουμε σήμερα. Η δουλειά που κάνατε είναι πραγματικά ε, πολύ μεγάλη. Δεν έχει τελειώσει βέβαια, είναι μακρύς ο δρόμος, αλλά επειδή είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής Μπαρόζο 1, πρέπει να σας πω ότι τα θέματα τα οποία εσείς θίξατε και προσεγγίσατε και, και οι μεταρρυθμίσεις που προτείνατε είναι τεράστια σημασία σε σχέση με αυτά που κάναμε εμείς τότε. Έτσι. Πρέπει να το πω αυτό και το λέω. Είναι καλό να το θυμίζουμε και δίκαιο. Ένα ερώτημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ζητάει από τα κράτη-μέλη, ε, ε, δεν τους τα θέτει πρώτων ευθυνών τους να πάρουν συγκεκριμένα δηλαδή μέτρα για μια φορολογική εναρμόνιση πολύ πιο προχωρημένη. Έτσι ώστε το σύνολο της Ένωσης να είναι ελκυστικό για τους ξένους με πραγματική νομική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παρέμβει στον τομέα τη άμεση φορολόγηση ω ένα επιπλέον στοιχείο της πολιτικής ελεύθερης κυκλοφορία, ε, είναι ένα θέμα συνέπεια των διαφόρων εργαλείων. Αν δεν θέλουμε οι δικηγόροι και οι διάφοροι σύμβουλοι να λένε στου πελάτε του να χρησιμοποιούν και να εκμεταλλεύονται τα κενά και τι φορολογικέ αποκλήσει, τότε πρέπει να πάψουν να υπάρχουν οι αποκλήσει. Οι νομοθεσίε των ίδιων των κρατών μελών δημιουργούν το forum shopping. Είναι ένα, ένα ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δεν είναι ζήτημα βέβαια απαθητικότητας της Κομισιόν. Η Κομισιόν πρέπει να, να φέρει το Συμβούλιο πρώτων ευθυνών του. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Μισελ, ο πρόεδρος. Ναι, Λουί, θα εξαρτηθεί από το πεδίο εφαρμογή ε, της φιλοδοξίας, το έβρος της φιλοδοξίας των κρατομελών. Να πάμε προ μια εναρμόνιση πλήρη εναρμόνιση, αν είναι αυτό το, αυτή η πρότασή σας, σε επίπεδο φορολόγησης των φυσικών προσώπων, ε, αυτή η φιλοδοξία είναι κάπως ακραία. Αλλά να σκεφτούμε πού στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε μια προσέγγιση στη, φορολογική, στη φορολογητέα βάση και στα ποσοστά, ε, αυτή είναι μια ιδέα την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε. Άλλωστε το φορολογικό ζήτημα αποφασίζεται με ομοφωνία, οπότε είναι δύσκολο να πάρθει οποιαδήποτε απόφαση ε, εκτός ε, εάν αλλάξει η συνθήκη. Στην επόμενη μετάθεση της συνθήκης θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθεί ε, ενισχυμένη πλειοψηφία ε, στο φορολογικό τομέα ή υπερενισχυμένη αν θέλετε, ιδάλλως δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσουμε. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η Περβάνς Μπέρες έχει το λόγο ε, για ένα λεπτό παρακαλώ κι εσείς. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, ήθελα να επανέλθω στο θέμα του καταλόγου των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει απορρίψει ήδη δύο φορές. Υπάρχει κάτι το παράδοξο εδώ. Όταν διαβάζει κανείς τον κατάλογο των χωρών ε, παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι ακόμα και στις χώρες ε, από τις οποίες η Κομισιόν ζητάει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μην παρέμβει Καϊμάν, Τζέρσι, Γκέρντζι, Βερμούδες, Παναμάς, Λίβανος. Ξέρω ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους φορολογικούς παραδείσους και τις χώρες που υπάρχει κίνδυνος ξελπνάτου χρήματος, αλλά είναι λεπτή αυτή η διαφορά. Ε. δηλαδή είναι λογικό να υπάρχουν υποψίες υπάρχει το ένα, ότι θα υπάρχει το ένα, θα υπάρχει και το άλλο. Τώρα κυρία Μύροβα, εντάξει, λέτε δεν μπαίνω εγώ στα χωράφια της και μπορεί να μην έχει τα μέσα στη διαθέση για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Η μονάδα πάντως που ασχολείται με τα μπόνους και με αυτούς τους κίνδυνους ξεπλήματος είναι μια μονάδα που αρχικά εξαρτώταν από τον Επίτροπο Χίλ και επειδή υπήρχε κίνδυνο σύγκρουση συμφερόντων μεταφέρθηκε προς την κυρία Γιούροβα. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να ήταν ε, όμως στην αρμοδιότητα του κυρίου Μοσκοβισή. Εάν λέμε ότι πρέπει να εξετάσουμε τις 200 χώρες, ε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό υπάρχουν χώρες για τις οποίες υπάρχουν υποψίες. Καλό θα ήταν λοιπόν να επικεντρωθούμε σε αυτές τις χώρες, να ξεκινήσουμε από αυτές. Τις ύποπτες χώρες και όχι να μιλάμε για έναν κατάλογο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ναι, σας είπα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επαναξετάσει τα ζητήματα στα οποία αναφερθήκατε προς το τέλος του έτους. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο σήμερα διότι οι αρμόδιοι επίτροποι αυτή τη στιγμή εξετάζουν λεπτομερώς τους μηχανισμούς. Βεβαίως αυτοί οι κατάλογοι θα συμπληρωθούν. Κατά τα λοιπά, επειδή αναφερθήκατε και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αύριο θα δείτε τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επί του ζητήματος. Θα τα δείτε αύριο αυτά. Το μέλλον είναι ήδη εδώ. Μάλιστα, Γιάννα Γκόμες, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας εξηγήσει τι έγινε στην εποχή της Τρόικας που, συμπεριέ, που συμπεριέλαβε ε, επί, ε, που έλαβε χώρα επί της εποχής Μπαρόσο. Είχαμε τεράστια φορολόγηση στην Πορτογαλία και τότε έφυγαν τα χρήματα στον Παναμά, παραδείγματος χάρη, στις offshore μέσω του, του, του, του ομίλου Σπύριτου Σάντου χωρίς κανείς να πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει σε παιδοκομισιόν Και είχαμε και τη φορολογική αμνηστία το 2012, έτσι. Η κομισιόν θα ασχοληθεί με το νέο σύστημα ξεπλήματος χρήματος που συμβαίνει σήμερα με τις χρυσές, θεω, χρυσές Visa Golden θεωρήσεις από διαβατηρίων. Συμβαίνει και στην ίδια χώρα μου ακόμα την Πορτογαλία και θα ασχοληθείτε επίσης με χώρες ε, με, με, το, με Freeport που υπάρχει και στη Λουξεμβούργο είναι μια νέα μορφή εξαλήματος χρήματος, έτσι. Και το οργανωμένο έγκλημα το χρησιμοποιεί αυτό, ακόμα και το η τρομοκρατία, για το Freeport μιλάω. Μάλιστα, ερωτήσεις ε, για το Freeport και για, As I said, previously. για τα αγορασμένα διαβατήρια, ναι. Ναι, υπάρχουν νέοι κανόνες για το καλό του χρήματος, για να αντιμετωπίσουμε κυρίως ε, την φοροαποφυγή αλλά και για την καταπολέμηση της, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτή η πρόταση εξετάζεται αυτή τη στιγμή, ξεκινήσει και τριμερής διάλογος με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οπότε τότε και εκεί θα συζητηθούν αυτά τα αισθήματα στα οποία αναφερθήκατε. Θα το εξετάσουν δηλαδή και τα άλλα θεσμικά όργανα για το Freeport δεν απαντάει ο κ. Γιούγκερ. Ναι, θα το εξετάσουμε το θέμα του Freeport, βεβαίως, λέει ο πρόεδρος. Ξέρω περί πρόκειται. Το έχουμε συζητήσει ήδη στο Λουξεμβούργο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, ε, ποπτείας του Λουξεμβούργου μου είπε ότι δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Το έχουμε ήδη ελέγξει λοιπόν. επόμενο, ο Άγγελ Τσαμπανσκή για το ECR. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, κύριε Πρόεδρε μάλλον της Επιτροπής, κύριε Γιούγκερ. Ε, έχουμε συζητήσει για τη φορολογία στο Λουξεμβούργο, τα Panama Papers, τις Ιρλανδικές περιπτώσεις και πραγματικά αυτό μας αναστατώνει όπως και να κάνει. Ας δούμε όμως προς το μέλλον. 1η Ιανουαρίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα. Ποια είναι τα μέτρα που σκέφτεστε να λάβετε έτσι ώστε να αποφύγουμε τα China Leaks. Τι θα κάνετε με τους Κινέζους εταίρους σας για το θέμα αυτό. Αγαπητές συνάδελφοι, από τις 15 ε, Νοεμβρίου του 2014 ως Κομισιόν προτείναμε ε, στο G20 να έχουμε ένα σύστημα αυτόματων ανταλλαγών πληροφοριών. Δεν συμφωνούσαν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι περισσότεροι διαφωνούσαν. Όμως ε, πάντοτε επανερχόμασταν σε αυτό το θέμα, στις διεθνείς ε, συναντήσεις, γιατί είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Έχουμε τους Τάμας Μάνα, Εύελιν Ρέγνερ και Έλλη Σλάιν. Ευχαριστώ πολύ, Ζαν Κλοντ. Πρέπει να πω ότι με εκπλήσει αλλά και χαίρομαι ότι παρά την κριτική που σου ασκήσανε, βλέπουμε ότι πολλοί είπαν ότι έχουμε ένα πρόεδρο επιτροπή, ο οποίο είναι δραστήριος, 12 πρωτοβουλίε. Ναι, ε, να υπάρχει ανταγωνισμός φορολογικός, αλλά να είναι πιο δίκαιος από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτό που ενοχλεί όμως είναι το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Μήπως λοιπόν ε, μπορούμε να πούμε στον πρόεδρο τη Επιτροπή ε, να μεταφέρει ότι πρέπει να σπάσει πια αυτή η ομοφωνία στο Συμβούλιο. Οι νομικοί λένε δεν γίνεται, αλλά πρέπει να ασκηθεί πολιτική πίεση. Ο Ζαν Κλοντ συμφωνεί μαζί μα ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Είπα στον Τόμας πριν από λίγα μόνο λεπτά ότι αν προκύψει θέμα ε, συνταγματικής ε, αλλαγής θα πρέπει να τεθεί το θέμα της ομοφωνίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από ειδική πλειοψηφία γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επόμενη, η Evelyn Ρίγνα. Ευχαριστώ πολύ. Πανέχομαι στα Freeports. Ε, αυτά που είπατε τίποτα δεν ήταν, επανέρχομαι. Free τι σημαίνει, σημαίνει δεν υπάρχει πόρος, δεν υπάρχουν δασμοί και πραγματικά είναι απίστευτο, απίστευτο το ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι δυνατόν ε, πολύτιμη λήθη ε, πίνακες, ε, πουθενά αυτά να μην φορολογούνται. Και είπατε ότι θέλετε λιγάκι να το δείτε. Η Κομισιόν όμως όταν θα διαπιστώσει ότι πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα, τότε τι θα κάνει, θα καταθέσει νομοθετικές προτάσεις, θα προσπαθήσει να ρυθμίσει το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πολιτική σημαίνει ρεαλισμός. Πριν κάνουμε κάτι πρέπει να το δούμε. Εγώ αυτό σας είπα, θα το δω. Σαφώς, πολύ σαφής λέει ο πρόεδρος, θα το δείτε λοιπόν, θα το αναλύσετε και ενδεχομένως θα πράξετε. Αυτό σημαίνει, να, βλέπετε τι σημαίνει η Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα πρωτοβουλίας και όχι το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γιούνκε, είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε, μια ανελαίτη, σε έναν ανελαίτητο φορολογικό ανταγωνισμό. Αρκεί να δει κανείς 0,005%. Υπάρχουν τέτοιοι φορολογικοί συντελεστές ε, στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Η Κομισιόν έχει κάνει τέλο πάντων κάποια πρόοδο, αλλά θα πρέπει να έχετε κατά νου ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μία πρόκληση που δεν μπορεί να λυθεί ούτε σε εθνικό ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αναπτυσσόμενε χώρε αυτέ πληρώνουν τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν country by country reporting που να είναι δημόσιο και θα φεύγει πέρα από τα όρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αφορά και το τι γίνεται στι τρίτε χώρε. Εδώ λοιπόν η Κομισιόν δεν κάνει τίποτα. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτές οι χώρες στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και ρωτώ συγκεκριμένα, η Κομισιόν τι θα κάνει για να αποφύγει εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ακριβώς διευκολύνουν τη φορολογική αποφυγή σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Και τι θα κάνει η Κομισιόν έτσι ώστε και αυτές οι χώρες να συμπεριληφθούν στην αναδιάταξη των φορολογικών μεταρρυθμίσεων. Ε, θα γίνει κάτι σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύει ο κύριος Γιούγκερ για αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ, Πρόεδρος της Επιτροπής. Ε, δεν ξέρω αν ε, καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέτε, ότι οι διεθνείς συμφωνίες οδηγούν στην φοροδιαφυγή. Εξαρτάται από τον τρόπο που εκτελούνται. Φυσικά οι αναπτυσσόμενες χώρες πλήττονται περισσότερο από άλλες και γι' αυτό το λόγο καταφέραμε να πείσουμε 85 χώρες ε, να συμμετάσχουν σε ένα σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ε, από όσο ξέρω, έτσι είναι. Θα σας δώσω συγκεκριμένες πληροφορίες όταν δω ακριβώ τη λίστα. Όμως το G20 καταφέραμε να πετύχουμε αυτό γιατί οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, ακριβώς πλήττονται περισσότερο και, επειδή κάποιες από αυτές υπάρχουν και, λαμβάνουν μέρος και στο G7, πραγματικά ασκήσαμε πίεση. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλα δύο λεπτά. Η κυρία Πιο Κορούνε Λέρνερ έχει το λόγο ως τελευταία για τη διαδικασία Catch the Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να υπάρχει συνοχή για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στην πολιτική ανάπτυξη παραδείγματος χάρη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Τράπεζα Ανοικοδόμησης συνεχώς χρησιμοποιούν ε, ταμεία επενδύσεων τα οποία είναι εγγεγραμμένα offshore και δεν έχουμε κάνει τίποτα γι' αυτό. Επίσης υπάρχει το θέμα των επιπτώσεων της φορολόγησης στις εμπορικές συμφωνίες μας. Πόσο, τι συγκεκριμένα κάνατε, το θέσατε το θέμα αυτό για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και τι θα κάνει η Κομισιόν στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής θα μπορούσε να μας πει κάτι γι' αυτό. Δεν κάνατε κάποια επερώτηση. Νομίζω ότι είναι η ίδια ερώτηση που έκανε και η κυρία Περβάνς για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Σε αυτό το θέμα πραγματικά παρακολουθούμε στενά το τι συμβαίνει. Αυτή ήταν η ερώτησή σας. Αυτή ήταν η απάντησή μου, δεν ξέρω όμως αν ήταν η ερώτησή σας. Ναι, αυτό ρώτησα, ναι. Ε, Εντάξει. Εδώ λοιπόν κλείνουμε. Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν μια ανοιχτή και δίκαιη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. 19 συνάδελφοι συνολικά έθεσαν ερωτήσεις. Πραγματικά σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Θα έχετε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή αυτών των δράσεων. Έχετε 15, έχουμε 15 λεπτά διάλειμμα.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

1, 2, tres. tres. continue Καλησπέρα. Συνεχίζουμε τώρα την ακρόασή μου. ω ε, προσκεκλημένο, θα μιλήσω τώρα την μετρική μου γλώσσα που είναι τα γερμανικά. ω ε, προσκεκλημένο έχουμε σήμερα τον ε, Υπουργό Φορολογικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, Φερνάντο Ρώσα Αντράντε. Ε, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντράδε που είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για την φορολογική κατάσταση στην Πορτογαλία και κάποια από τα νησιά σας. Στο τέλος της συζήτησής μας με τον πρόεδρο Γιούνκερ αναφέρθηκε και το ζήτημα της Μαδέιρα. Σήμερα θα έχουμε σίγουρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Όπως είναι φυσιολογικό, έχουμε 45 λεπτά, όπως κάνουμε συνήθως, και κανονικά έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, ένα λεπτό η ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση. Ξεκινάμε λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Έχετε αμέσως ε, το λόγο για την εισαγωγή που, θα, που έχει προβλεφθεί για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε να μιλήσω σε αυτήν εδώ την Ειδική Εξεταστική Επιτροπή. Θα ξεκινήσω τονίζοντας τη σημασία του θέματος ε, και τη δουλειά που η Επιτροπή έχει ε, καταφέρει να φέρει εις πέρα στα τελευταία χρόνια για τους φορολογικούς ε, παραδείσους ε, που χρησιμοποιούν διάφοροι για να κρύψουν τον πλούτο τους από τις δημόσιες υπηρεσίες επίσης για να κρύψουν τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες. Αυτές οι πρακτικές ε, δεν υποσκάπτουν μόνο τα φορολογικά έσοδα, αλλά και γενικότερα την ομιμότητα των φορολογικών συστημάτων. Οι αποκαλύψεις ε, μέσω των Panama Papers οδήγησαν την κοινή γνώμη στο να δώσει προσοχή για άλλη μια φορά σε αυτό το θέμα, στις διάφορες πρακτικές ε, φοροδιαφυγής. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, οι δικές μας αρχές, όπως και οι αρχές άλλων χωρών, βρήκαν τα άτομα που αναφέρονται στα Panama Papers. 165 κάτοικοι της Πορτογαλίας αναφέρονται στα Panama Papers και είναι τώρα υπό διερεύνηση. Η ομάδα εργασίας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική ε, στα πλαίσια του ΩΣΑ και στο ειδικό φόρουμ GSIC. Έχουμε μάθει κάποια πράγματα όμως από αυτές τις αποκαλύψεις. Οι πληροφορίες που αποκάλυψαν τα Panama Papers ε, μας ε, δίνουν κάποια στοιχεία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε την έρευνά μας. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι αυτά τα στοιχεία θα μας δώσουν και νέες μεθόδους για να μπορέσουμε να βρούμε πληροφορίες, γιατί αυτές που έχουμε σε πολλές περιπτώσεις είναι ανεπαρκείς. Δημοψιοποιούνται με γεγονότα, αλλά είναι πολλές φορές ε, παλιά, παροχημένα και σε πολλές περιπτώσεις οι σχέσεις μεταξύ ατόμων και χωρών δεν έχουν κάποιο νόημα για φορολογικούς σκοπούς. Η αυτόματη όμως ανταλλαγή πληροφοριών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιδράσουμε σε μια τέτοια κατάσταση και προληπτικά. Γι' αυτό το λόγο, μέσα από την Εθνική Νομοθεσία της η Πορτογαλία έχει λάβει πρωτοβουλίες σε διμερές και πολυμερές επίπεδο υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και πιο ενδελεχής. Η πρόσκληση που μου στείλατε ανέφερε τις μεταφορές σε τοποθεσίες με προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα. Στην Πορτογαλία υπάρχει μια τέτοια μορφή μεταφορών συν η υποχρέωση ε, να, να, να δημοσιοποιούνται οι στατιστικές. Μεταξύ του 2000-2014 είδαμε ότι τα δεδομένα δεν ήταν σωστά σε επίπεδο στατιστικής και διαρευνούμε την ρίζα αυτού του προβλήματος. Υπάρχει όμως ένα σχόλιο εδώ, ένα σύστημα που ελέγχει τις μεταφορές ε, χρημάτων ε, είναι ευάλωτο στις τριγωνικές συναλλαγές. Αν γίνει η μεταφορά σε μια ενδιάμεση χώρα που δεν έχει σύνδεση με την χώρα που διεξάγει τη συναλλαγή, θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί η διαδρομή της συναλλαγής. Διότι ο χώρος, η χώρα κατοικίας δεν μπορεί να διαπιστώσει ότι τα χρήματα δρομολογούνται προς ένα φορολογικό παράδεισο. Γι' αυτό χρειάζεται ένας μηχανισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών. Έτσι ώστε να μπορούν ε, όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δίνουν τις πληροφορίες που απαιτεί ας πούμε, η πορτογαλική κυβέρνηση αλλά και το κάθε κράτος μέλος να μπορεί να γνωρίζει για κάθε μεταφορά χρημάτων ή συναλλαγή που πηγαίνει από τη μία χώρα στην άλλη μέσω ενδιάμεσων. Γι' αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσουν οι ευρωπαϊκές πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που ήσασταν ε, έτοιμος να έρθετε εδώ στις Βρυξέλλες. Θα κάνουμε και μία αποστολή για fact-finding mission στην Πορτογαλία και θα δούμε περισσότερα πράγματα. Δίνω ε, το λόγο στους ε, εισηγητές τώρα. Ο κύριος Καφόντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή να εξηγήσετε την κατάσταση στην Πορτογαλία. Είμαι περίεργο σε σχέση με αυτό που αναφέρατε για τις μεταφορές που δεν εποπτεύονται από το 2011 στο 2014. Ε, μίλησατε για δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Μπορείτε να μας πείτε πώς συνέβη αυτό, πώς είναι δυνατόν να, να πάνε σε φορολογικές παραδείσεις τόσα πολλά χρήματα χωρίς καμία εποπτεία και ποιοι ήταν οι δικαιούχοι, ποιοι είναι οι φορολογούμενοι, ποιοι είναι οι μεσάζοντες. Πολλές φορές αναφέρεται η Τράπεζα της Πορτογαλίας ε, ως μεσάζοντας. Μπάνκο του Πορτογάλ. Και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Ο εισαγγελέα που εξετάζει το εξέτημα χρήματος ε, ε, έχει επαρκή πρόσβαση, υπάρχει επαρκή συνεργασία από τις φορολογικέ αρχέ στην Πορτογαλία. Λαμβάνει όλες τι πληροφορίε που χρειάζεται για να κάνει την έρευνά του. Και επειδή ήσασταν υπό την εποπτεία της Τρόικα, ε, τι ρόλο έπαιξε η Τρόικα για να προλάβει αυτή τη μαζική και ανεξέλεγκτη μεταφορά χρημάτων προς ορολογικούς παραδόσεις ε, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά αυτές τις μεταφορές τις ανεξέλεγκτες, από όσο γνωρίζουμε, η οι χρηματοοικονομικοί όμιλοι έκαναν τη δουλειά τους, έστειλαν τα στοιχεία δηλαδή στις φορολογικές αρχές, όμως η επεξεργασία των δεδομένων στο επίπεδο των, οικονομικών αρχών ε, για συναλλαγές ε, ύψους 10 δισεκατομμύριων ευρώ δεν έλαβαν χώρα. Δεν έλαβε χώρα επεξεργασία, δεν συμπελήθηκαν στη βάση δεδομένων, στη βάση δεδομένων δεν είχε γίνει επεξεργασία δεδομένων και δεν πήγαν στα στατιστικά στοιχεία. Ούτε προσθέθησαν ε, ε, σε κάποιο πλαίσιο επιθεώρησης, ε, ούτε εντάχθηκαν σε κάποιο πλαίσιο. Οι φορολογικές αρχές τώρα έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα. Είπα λοιπόν, οι τράπεζες είχαν στείλει τα δεδομένα, αλλά δεν είχε γίνει επεξεργασία τους από τις αρχές. Ο εισαγγελέα στη χώρα μου έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ποινική για αυτήν την ε, αποτυχία, αν θέλετε. Θα υπάρχει πρόσβαση, λοιπόν, πλέον και για το μέλλον. Δεν υπήρξε πάντως παρέμβαση ε, της Τρόικας ό,τι αφορά τη μεταφορά χρημάτων ε, προς τις offshore. Ο Πίτερ Γιάτσεκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Υφυπουργό που είναι εδώ μαζί μας ε, θα ήθελα να ξέρω πώς αξιολογείτε την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, της σχετικής στη χώρα σας. Ο πρόεδρος της Επιτροπής ήταν εδώ προηγουμένως, ο κύριος Γιούνκερ. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, πώς πάει. Ποιο είναι το επίπεδο διάδρασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι γίνεται με την εφαρμογή ε, της νομοθεσίας στη χώρα σας. Η εποπτεία όλων των μεσασόρων και όχι μόνο των τραπεζών, των δικηγόρων, ε, των ε, φορολογικών συμβούλων, ε, πώς πάει στη χώρα σας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. για το ρόλο των θεσμικών οργάνων. Ήταν ε, θεμελιώδης για τη θέσπιση του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών. Να πω, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική αλλαγή ε, στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές πλαίσιο πλέον. Θα έχουμε πρόσβαση ε, σε πληροφορίες από ξένες δικαιοδοσίες, από ξένα δικαιοδοτικά όργανα. Ε, δεν είναι πια τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσοστό φορολόγηση της κάθε χώρας, εφόσον η χώρα αυτή όμως δίνει τις πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία ε, σε ό,τι αφορά το, τα κέρδη τα οποία ε, προκύπτουν στο έδαφος μιας χώρας να φορολογείται εκεί δηλαδή, να φορολογείται εκεί αυτά τα κέρδη. Εμείς έχουμε λάβει υπόψη μα τι συστάσεις του ΩΣΑ. Ε, πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Οι μηχανισμοί εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα ε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό που υπάρχει είναι η ανταλλαγή πληροφοριών. Και η εφαρμογή της ε, φορολογικής νομοθεσίας είναι πρωτίστως θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο. Να δημιουργήσουμε δηλαδή μηχανισμούς που να επιτρέπουν στις εθνικές φορολογικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ήσασταν ακριβείς στο χρόνο σας, αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα, ο κύριος Μέλος, πρώτος εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινάτε να μετράτε το χρόνο της ερώτησής μου, πριν ξεκινήσει η ερώτησή μου, παρακαλώ σταματήστε το ρολόι. Ήθελα να θέσω ένα ζήτημα για αυτή τη συζήτηση. Είναι πολιτική, αλλά πρέπει να βασίζεται σε γεγονότα, όχι έτσι σε γενικές αναφορές. Έκανε μια ερώτηση ο κύριος Κόφοντ, ο εισηγητής από την ομάδα των σοσιαλιστών. Να σας ενημερώσω εδώ, εκεί στο πανέλ ότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε 10 δις ε, μεταφορές που δεν καταγράφηκαν μεταξύ του 2011 και του 2014. Δεν πρέπει να υπάρχει παρεξήγηση εδώ. Δεν έχει σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει η κυβέρνηση. Ο Γενικός Διευθυντής ε, για τις φορολογικές επιθεω... επιθεωρήσεις αναφέρθηκε στις ε, φορολογικές δηλώσεις που έγιναν την περίοδο 2015-2016 και αυτές, ε, τέσσερις από αυτές ήταν όταν υπήρχε η τερέχουσα κυβέρνηση. 18 από 20 λοιπόν από τις ε, ε, εκθέσεις ε, ήταν σε αυτό το διάστημα 20 εκθέσεις, ε, οι τέσσερις 4 υπό την τρέχουσα κυβέρνηση. Τώρα μπορώ να ξεκινήσω με την ερώτησή μου. Να σας καλωσορίσω και να σας μιλήσω τώρα για μια μυστική συμφωνία που επιβεβαιώθηκε στις 28 Αυγούστου του 2010 μεταξύ του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Πορτογαλίας και του Πρωθυπουργού, του κυρίου Σόκρατες. Συμφωνήθηκε ότι ο Παναμά θα, Παναμάς θα βγει από τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία λοιπόν έκανε τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να βγει ο Παναμάς από τον κατάλογο. Τελικά όμως ο Παναμάς παρέμεινε στον κατάλογο χάρη στις πρωτοβουλίες του Σοσιαλιστικού Κόμματος ε, της Πορτογαλίας του PSD, συγγνώμη, των Σοσιαλδημοκρατών της Πορτογαλίας. Ε, αν θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε την ε, νομοθεσία για τους φορολογικούς παραδείσους, η Ουρουγουάη και άλλες χώρες αναφέρεται ότι πρέπει να βγουν από την λίστα. Όμως αυτό δεν ακολουθεί τα κριτήρια αβγ του άρθρου 362D. Ε, τελικά, τι έχετε να πείτε για μια κυβερνητική απόφαση η οποία τελικά παραβιάζει ε, την νομοθεσία. Μπορεί, δεν μπορεί να παραβιάζει την νομοθεσία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Και κύριε Υπουργέ, θα καταλήξω τώρα γι' αυτά τα δέκα δις ευρώ. Κάποιες από αυτές τις ε, μεταφορές έγιναν όταν ήσασταν εσείς κυβέρνηση. Ποιος έλαβε μέρος, ποιες ήταν οι τράπεζες, πώς έγινε. Ε, πρέπει ε, να απαντήσετε σε πολύ λίγο χρόνο, αν τηρήσουμε το χρόνο, οπότε σας δίνουμε περισσότερο χρόνο για την απάντησή σας. Παρακαλώ. Αξιότιμε κύριε Μέλο. Δεν πρόκειται να διορθώσω τα νούμερα που μου θέσατε. Όμως υπάρχουν νομικά σφάλματα που έχουν να κάνουν με το επαγγελματικό απόρριτο, το τραπεζικό απόρριτο κτλ. Πολλές φορές ε, με αμέλεια αντιμετωπίστηκαν αυτά τα ζητήματα. Τώρα για τα ερωτήματα που θέσατε. Άκουσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι δεν ήμουν μέλος σε καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που αναφέρατε ότι σε δύο περιπτώσεις ο πρωθυπουργός της χώρας μου και ένας άλλος πρωθυπουργός ε, μιας χώρας ε, η οποία κυβερνεί από το δικό σας κόμμα ε, ζήτησαν να βγει ο Παναμάς από τους φορολογικούς παραδείσους το 2010. Επίσης, Αναφέρθηκε ο ότι ο κύριος Πάσος Κοέλιο, ο Πρωθυπουργό, επισκέφθηκε τον Παναμά. Όμως εγώ απαντήσεις μπορώ να δώσω μόνο εκ μέρους της δικής μας κυβέρνησης. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση στον κατάλογο αυτό, διότι αυτό που εμείς τις αποκαλούμε δεν είναι φορολογική παράδειση, αλλά μη συνεργαζόμενες δικαιοδοσίες γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στις φορολογικές πληροφορίες. Ε, το σημαντικό δεν είναι ποιοι είναι οι φορολογικοί συντελεστές στην κάθε χώρα, το θέμα είναι η διαφάνεια. Η απόφαση κυβερνητική που αναφέρατε ήθελε να βγάλει τρεις χώρες από τον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων που είναι μεγαλύτερος από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή ε, χώρα. Τρεις λοιπόν ήταν οι χώρες που βγήκαν γιατί πληρούσαν μια σειρά κριτηρίων. Αντάλλαξαν δηλαδή πληροφορίες με την Πορτογαλία μέσω μηχανισμών που δεν τίθενται από τις διεθνείς συνθήκες αλλά είναι αποδεκτές από τον ΟΣΑ ως μέσο ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτά τα κριτήρια στην ουσία δεν έδιναν τη δυνατότητα στην Πορτογαλία να βγάλει τον Παναμά από, το, από τη λίστα και αυτό το είπαμε ξεκάθαρα στον πρέσβη του Παναμά. Η κυβέρνηση αυτή λοιπόν δεν θέλει σε καμία περίπτωση να υπάρχει κάποια συγκάλυψη ε, σε επίπεδο διεθνών συναλλαγών και σχέσεων. Το λέω ξεκάθαρα. Τώρα για την προηγούμενη κυβέρνηση, η δική μας κυβέρνηση διόρθωσε μια κατάσταση ε, κατά την οποία οι στατιστικές για τις μεταφορές ε, χρημάτων ήταν ε, λανθασμένες. Πρόκειται για δημόσια στοιχεία. Τα δεδομένα που δημοσιεύονται, που δεν δημοσιεύονται, δεν δημοσιεύονται όχι επειδή είναι απόρριτα, αλλά επειδή η νομοθεσία της Πορτογαλίας ε, ορίζει ότι είναι θέμα φορολογικού απορρίτου όπως για όλους τους πολίτες. Μια σύντομη επερώτηση. Πολύ σύντομη. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ε, αναφέρω τον νόμο 63D της φορολογικής νομοθεσίας και θα σας πω και ακριβώς ε, όλες, ε, ε, όλη τη διατύπωσή του. Και μετά θα μας πείτε εάν η Πορτογαλία έχει, συμμορφώνεται με την νομοθεσία για τους φορολογικούς παραδείσους ή όχι, συγγνώμη, 68. 80 και 81 είναι τα άρθρα, τα σχετικά. Ναι, στείλτε τα στη γραμματεία αυτά τα στοιχεία για να προχωρήσουμε παρακαλώ. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα ελέγξουμε τις πληροφορίες. Επόμενη μιλήτρια η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Αναρωτιέμαι γιατί υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Ποια είναι η αιτιολόγηση για να καθυστερήσει η έρευνα ε, την οποία έχετε ζητήσει για την περίοδο 2011-2014. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν τι συνέβη μετά το 2015, το 2016, όταν πια είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας. Ήθελα λοιπόν να ξέρω εάν αυτές οι μεταβιβάσεις, οι οποίες ερευνώνται αυτή τη στιγμή, περιλαμβάνουν και τη Μαδέιρα. Και γιατί πόσα μιλάμε. από και προς τη, και Μαδέρα κυρίως ε, το 2015. Ήθελα επίσης να σας ρωτήσω για την, ε, τις δικαιοδοσίες ε, ε των μεσαζόντων που εμπλέκονται. Περιλαμβάνονται χώρες όπως η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο. Μιλάμε για οικονομικά κέντρα στα οποία στέλνουν οι Πορτογάλοι συχνά τα χρήματά τους. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος ε, και στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες, ό,τι αφορά την απάτη ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, και πόσα από αυτά περνούν από το λιμάνι του Ρότερνταμ. Ο κύριος υπουργό έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ αξιότιμο μέλος. Ε, η έρευνα στην οποία αναφερθήκατε διενεργείται από διάφορα σώματα του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουμε ακόμα την τελική έκθεση. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, οπότε αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι κάνουμε εμείς εν το μεταξύ, ακούστε, αυτό είναι ένα ζήτημα πληροφορική στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε κάποια ένδειξη αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα μεταξύ 2013 και 2016. Το 2016 το εντοπίσαμε, από όσο γνωρίζουμε. Δεν πρόκειται για κάτι ε, σημαντικό, κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Τώρα, η Μαδέιρα είναι, αποτελεί μέρος της Πορτογαλίας, έτσι είναι πορτογαλικό έδαφος. Έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώ βέβαια. Οι κανόνε που ισχύουν πάνω στην Πορτογαλία ισχύουν και στη Μαζέιρα. Δεν υπάρχουν χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι σε μαύρο κατάλογο, διότι ε, είναι κατά τη πορτογαλική νομοθεσία. Παρακαλώ, επόμενο ομιλητής. Όχι, η κυρία Γκόμες επανέρχεται. Έχουμε την πληροφορία ότι ο Γενικός Διευθυντής ε, των ε, Επιθεωρητών έχει κλείσει την έρευνα αυτή. Μπορεί να μην έχει λάβει ακόμα την έκθεση, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τελικά τι συμβαίνει. Επίσης, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ, όταν συζητήσατε το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο, αναφερθήκατε στο γεγονό ότι 97% των μεταφορών, των μεταβιβάσεων αυτών, αφορούσαν ε, τον τροπεζικό όμιλο BES που έχει καταρρεύσει έκτοτε. Έχετε κάτι να πείτε από αυτού. Ναι, συγγνώμη, για λόγους που εξήγησα και στον κύριο Νούνος, Νούνες Μάλλο, ε, εγώ σεβόμενος στην προγραμματική νομοθεσία δεν μπορώ να σας δώσω ε, τα ονόματα των χρηματοπιστατικών ομίλων που ε, διέπρεξαν αυτές τις μεταφορές. Τα στοιχεία τα οποία είναι δημόσια, έχουν να κάνουν με την χώρα ε, προορισμού. Αυτά μπορείτε να βρείτε και στο ίντερνετ. Δεν λέμε όμως ποια, ποιος είναι ο τραπεζικός όμιλος ε, προέλευσης. Οπότε μπορώ να σας δώσω την πληροφορία. Λοιπόν, οι δύο μεγάλες ε, πολιτικές ομάδες εξάντλησαν το χρόνο τους. Ε, πάμε τώρα στην πολιτική ομάδα ECR. η Πορτογαλία βρίσκεται υπό πρόγραμμα ε, πρόγραμμα που συνεργάζονται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τι έχετε λοιπόν συζητήσει για την Μαδέρα, για το χρηματοψηφιακό τομέα και ποιες είναι οι προσπάθειες ε, κατά της ε, φοροαποφυγής ε, στην Πορτογαλία. Αυτές νομίζω ότι είναι προτεραιότητες για τους πιστωτές. Και πώς ακριβώς συζητήθηκαν λοιπόν τα θέματα αυτά. Ο κύριος Υφυπουργός έχει το λόγο. Νομίζω ότι εδώ πρόκειται για δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Αφενός γίνεται αναφορά στο φορολογικό σύστημα στη Μαδέιρα, αυτό το ειδικό καθεστώς ε, στο ελεύθερο λιμάνι της Μαδέιρα όπως αποκαλείται. Αυτό το φορολογικό καθεστώς ε, θεσπίστηκε ε, στο πλαίσιο ενός κανονισμού όπου θέλαμε να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη των, οικονομικών, των εξόχως απομακρυσμένων περιοχών. Πρόκειται λοιπόν για υποστήριξη τη της ε, Μαδέρα και εδώ και κάποια χρόνια όμως ε, πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν πια διατάξεις ε, για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτό το θέμα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών νομίζω πλέον ανήκει στο παρελθόν. Πάω τώρα στο θέμα της ε, αντιμετώπισης της ε, φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. Αναμφίβολα, αυτό ήταν προτεραιότητα πολλών ε, κυβερνήσεων. Αυτό το έδειξε και η κυρία Γκόμες. Πρόκειται, παραδείγματο χάρη για το θέμα του ΦΠΑ ή για το γεγονός ότι τα ποσά ΦΠΑ ήταν υποτιμημένα Άλλο θέμα που τίθεται επιτάπητος είναι το θέμα των περιουσιακών στοιχείων. Στην Πορτογαλία λοιπόν προσπαθήσαμε να συστήσουμε κάποιους ε, μηχανισμούς και σε μεγάλο βαθμό ε, ακολουθήσαμε τις οδηγίες ε, του μηχανισμού BEPS. Αλλά έχουμε κατά νου και άλλους μηχανισμούς, παραδείγματος χάρη την άρση της δυνατότητας να διακυβεύονται μόνο κάποια μικρά ποσά. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα όπου προσαρμόσαμε τη νομοθεσία με στόχο να επικρατεί διαφάνεια στο χρηματοψηφιστικό τομέα ή να καταπολεμηθεί το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Ο κύριος Βέγκας από την ΚΟΕ. Κοιτάξτε, ε, μία σύντομη ερώτηση προς εσάς. Αφενός ε, πρόκειται για το θέμα το, της έρευνας ε, για τα Panama Papers αλλά και για τα Swiss Leaks όπου επίσης διαπιστώθηκε ότι φύγονται 611 φορολογούμενοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα άτομα αλλά ο απολογισμός. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση και τελικά τι εισπράξατε. μπορέσατε να μειώσετε τη ζημιά από τη φοροδιαφυγή. Και νομίζω ότι αυτή την πληροφορία πρέπει να την δημοσιοποιήσετε. Επίσης, σε το θέμα του τραπεζικού και φορολογικού απορρίτου. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν τι σημαίνει αυτό σήμερα και πώς αντιμετωπίζετε σήμερα ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η φοροδιαφυγή. Εξάλλου, ε, τι μέσα έχετε στη διάθεσή σας για να αντιμετωπίσετε τις νέες προκλήσεις, ε, τις νέες διατάξεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι είδου απαντήσεις ε, μπορείτε να δώσετε οποτεδήποτε τίθενται επιτάπητε σε αυτά τα θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής. Και μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Συστάσεις αναχώρα. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα αυτό και γνωρίζω ότι στην Πορτογαλία προβλέπεται τα αποτελέσματα να υποβάλλονται αναχώρα. Στην Πορτογαλία όμως ε, το κατώτατο όριο είναι υψηλότερο, 750 εκατομμύρια ευρώ λοιπόν, πριν μεταφερθούν τα στοιχεία. Εμείς εδώ στο Κοινοβουλίο μιλάμε για το κατώτατο όριο και θα θέλαμε να ξέρουμε πόσες εταιρείε εμπίπτουν και είναι πάνω μάλλον από αυτό το όριο, τα 750 εκατομμύρια και καλύπτονται από τις σχετικές διατάξεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Όσον αφορά τα Swiss Leaks και τα Panama Papers, μπορώ να σας πω ότι οι περισσότερες ε, πληροφορίες ε, που περιλαμβάνονται στα έγγραφα είναι πλέον απαρχαιωμένες, ξεπερασμένες. Είναι πολύ δύσκολο να εισπράξει κανείς ε, φόρους, μάλιστα οι αρμόδιες αρχές εν μέρη δρομολόγησαν και ποινικές ε, διαδικασίες. Υπήρξαν καταστάσεις ε, από το 2004 μέχρι το 2006. Εντοπίστηκαν αυτές οι περιπτώσεις ε, επειδή όμως προχώρησαν και αργότερα, ε, γι' αυτό συνεχίζεται η διαδικασία. Όσον αφορά τα Panama Papers, ξεκινήσαμε τις έρευνες πριν από κάποια χρόνια. Τώρα εξακολουθούμε να ερευνούμε τα περισσότερα έγγραφα για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εισπράξουμε κάποια πρόστιμα. Αλλά είναι αλήθεια ότι Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απορρέουν όμως από διαρροές. Αυτό που έχει σημασία είναι ε, να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε με επίσημη ανταλλαγή πληροφοριών. Και γι' αυτό το λόγο ενισχύσαμε και την ε, πληροφορική και το ανθρώπινο δυναμικό μας. Είναι πολύ δύσκολο για μια μικρή χώρα να επεξεργαστεί όλη αυτή την πληθώρα των πληροφοριών. Όσον αφορά το κατόφλι ε, που αναφέρεται στις ε, αναχώρα στάσεις, θέλω να σας πω ότι όταν ορίζει κανείς ένα κατώτατο όριο, ε, προφανώς και ενδιαφέρουν και στοιχεία που έρχονται από άλλες χώρες. Για το θέμα δεν είναι να βάλει κανείς τόριο στη δική του τη χώρα. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η Πορτογαλία ενδιαφέρεται το όριο να ορίζεται συλλογικά, αλλά όπως και σε άλλες χώρες, κατ' ουσίαν καμία χώρα τώρα ε, δεν αισθάνεται το κίνητρο να ε, φορολογείς περισσότερο εταιρείε που βρίσκονται στη δική της την επικράτεια σε σχέση με άλλες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν είναι απλά απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις ε, διάφορες χώρες. Δύο ακόμα θέλουν να ζητήσουν το λόγο. Γκίγκολ και Φερνάντες. Σφέν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Χαοτική τη βρίσκω σήμερα mm τη διαδικασία. Αυτό πρέπει να σας το πω. Θα μιλήσω τώρα αγγλικά. Τρία, πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Μετά τις αποκαλύψεις, εσείς θεωρείτε ότι υπήρξε παραβίαση των υποχρεώσεων περί ξεπλήματος χρήματος από την Πορτογαλία, διότι τα στατιστικά στοιχεία για τις διασυνοριακές μεταφορές κεφαλαίων δεν δημοσιεύθηκαν στο παρελθόν όπως προβλεπόταν. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Έχετε αποφασίσει να παρακολουθήσετε τις τράπεζες εκείνες ιδιαίτερα που δεν είχαν ελεγχθεί στο παρελθόν και που εμπλέκονται στα Panama Papers. Και έχετε ξεκινήσει ε, διαδικασία δίωξης κατά των τραπεζών αυτών. Και ποιος εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του ξυπνήματος χρήματο εφαρμόζονται. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να διευκρινιστεί για να εξασφαλίσουμε ότι οι υποχρεώσεις εφαρμόζονται όντως. Ευχαριστώ. Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ακούστε, να διευκρινίσω καταρχήν ένα πράγμα. Οι υποχρεώσεις τις οποίες αναφέρθηκα είναι υποχρεώσεις που υπάρχουν μόνο σε επίπεδο φορολόγησης. Είναι κάτι ξεχωριστό δηλαδή από το σύστημα ελέγχων που έχουν να κάνουν το ξέπλυμα χρήματος. Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στην Πορτογαλία, η αναφορά που πρέπει να δίνεται για τις μεταβιβάσεις από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς πρέπει να περνούν από την νομοθεσία ξεπλήματο χρήματο. ε, σύμφωνα με την νομοθεσία πάνε προς την κεντρική τάξη τη Πορτογαλίας και όχι προς τις εθνικέ αρχές. Είναι διαφορετικά συστήματα αυτά. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχουν ζητήματα που να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος σε αυτή την περίπτωση. Το EFTF επισκέφθηκε την Πορτογαλία πριν από λίγο. Θα έχουμε λοιπόν μια πιο ανεξάρτητη αξιολόγηση σε λίγο καιρό. Όμως η εντύπωση που έχω εγώ είναι ότι το σύστημα ελέγχου στην Πορτογαλία βασίζεται σε αναφορά προς την Τράπεζα της Πορτογαλίας, την Κεντρική Τράπεζα της Πορτογαλίας. Και βεβαίως υπόκειται σε έλεγχο από την αστυνομία και από ε, την εισαγγελία. Αυτό είναι το σύστημα, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε για τις φορολογικές διοικήσεις, βεβαίως όποτε ε, υπάρχει κάποια παράβαση αυτή τη χάνει αναφοράς προς τις δικαστικές αρχές, από τις φορολογικές αρχές δεν νομίζω να υπάρχει οποιαδήποτε επέμβαση εδώ του Υπουργείου. Οι πληροφορίε που έχω εγώ στη διάθεσή μου είναι ότι η πρόθεση, ε, μάλλον δίνεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή σήμερα σε αυτές τις οργανώσεις και αυτά τα πρόσωπα, νομικά και φυσικά, τα οποία κάνουν αυτές τις δύο συναλλαγές. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες σχόλια. Έχουμε εδώ κάποιους ε, κανόνες, κύριε συνάδελφε. Ε, να πω ότι εκπλήσωμαι γιατί παραβιάσεις και τα φορολογικά εγκλήματα θα πρέπει να είναι να προηγούνται της ξεπλήματος του χρήματος ως αδίκημα. Το να τα διαχωρίζετε μου φαίνεται περίεργο. Μπορείτε να μας πείτε γιατί αυτές οι δύο πλευρές δεν συνεργάζονται. Επίσης, όταν έχετε ευρήματα για το ξέπλυμα χρήματος, θα πρέπει να πηγαίνει στην εποπτική αρχή τραπεζών η πληροφόρηση φυσικά, για να υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία. Με την απάντησή σας, στην ουσία, φαίνεται ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ε, ε αρμόδιων οργάνων. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ήμουν αρκετά ξεκάθαρος. Να ξεκαθαρίσω τώρα την απάντησή μου. Το όλο σύστημα ελέγχου το, του ξεπλήματος ε, μαύρου χρήματος βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχουν λοιπόν ενημερώσεις από την τράπεζα στις εποπτικές αρχές, που είναι η ε, τράπεζα της Πορτογαλίας. Και αυτό αυτή η κοινοποίηση είναι κάτι στο οποίο έχει πρόσβαση το δικαστικό σύστημα. Ε, έχουμε πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όταν μιλάμε για ύποπτες συναλλαγές. Οι μεταφορές χρημάτων στις offshore έχουν άλλο στόχο. Είναι φορολογικός και όχι ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Φυσικά οι φορολογικές αρχές ε, λαμβάνουν μέρος στο σύστημα κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Όμως οι φορολογικές αρχές αν ανοιχνεύσουν κάποια εγκληματική δραστηριότητα ή υποπτή δραστηριότητα. Ειδικά ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε θα το παρακολουθήσουν. Αν υπάρχει υποψία δηλαδή για το έγκλημα ξεπλήματος μαύρου χρήματος ε, ε ως προς οποιαδήποτε συναλλαγή offshore ε, που ανοιχνεύουν οι φορολογικές αρχές, απαραίτητα τα στοιχεία δίνονται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, έτσι ώστε να ε, μπορέσει να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο ο συνάδελφος Χωσέ Μανουέλ Φερνάνδες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν ε, δύο μέρη στην ερώτησή μου, ε, η οποία στην πρώτο μέρος θα έχει απάντηση ναι ή όχι κατά πάσα πιθανότητα. Το κάνετε με τον κύριο Μάλλο. Η πορτογαλική κυβέρνηση έβγαλε τρεις χώρες από την λίστα με τους φορολογικούς ε, παραδείσους. Το ζήτησε η κυβέρνηση από τις φορολογικές αρχές αυτό. Οι φορολογικές αρχές έλαβαν μέρος στην όλη διαδικασία και τις ακούσαμε προσεκτικά κατά τη θέσπιση των κανόνων. Υπήρξε μια σειρά γνωμοδοτήσεων που έδωσαν οι φορολογικές αρχές και πλέξαν πλήρως στη διαδικασία. Οπότε να βγάλω το συμπέρασμα κύριε Υπουργέ ότι οι φορολογικές αρχές ε, ε, γνωμοδότησαν θετικά ως προς αυτό. Δηλαδή, ε, αν αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο του διατάγματος στάλει στο κέντρο φορολογικών μελετών και ε, από εκεί πήραμε το πράσινο φως, όχι δεν έγινε έτσι διαδικασία. Οπότε να συμπεράνω το αντίθετο, ότι δεν έδωσαν θετική γνωμοδότηση οι φορολογικές αρχές. Τις πληροφορίες σας τις έδωσα. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να συμπεράνετε. Οπότε ε, συμπεραίνω ότι δεν υπήρχε θετική γνωμοδότηση από τις φορολογικές αρχές. Ωραία. Δεν βλέπω κάποια άλλη ερώτηση. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Υπουργό. Σε τρεις ή μισή εβδομάδες έχουμε μία αποστολή fact-finding στην Πορτογαλία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και με αυτήν την ευχαρίστηση, με αυτή την ευχαριστία να κλείσω τη σημερινή συνεδρίαση. Όταν έρθουμε στην Πορτογαλία θα συνεχίσουμε πιο εντελώς τη συζήτησή μας. Ε, κλείνουμε τώρα την συνεδρίαση της ομάδας και μετά έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών που δεν είναι δημόσια. Παρακαλώ στο μεταξύ όσοι δεν έχουν δικαίωμα να είναι εδώ στην συνεδρίαση και κλεισμένων των θηρών να φύγουν. Ευχαριστώ.